Uh, uh, Να καλωσορίσω θερμά όλους ε, το απόγευμα. Συγγνώμη που ξεκινούμε ελαφρώς αργότερα. Στο γεύμα υπήρχε μια συνάντηση. Να σας καλωσορίσω στην τελευταία συνάντηση για το 2013, η οποία λαμβάνει χώρα σήμερα και αύριο. Έχουμε πολλές προτάσεις με αρκετές λεπτομέρειες που θα πρέπει να συζητήσουμε και κάποια σημαντικά αύριο, τα οποία ξέρω ότι θα ενδιαφέρουν όλους σας. Οπότε να σας υπενθυμίσω απλώς ότι η ψηφοφορία θα έχουμε από τις 9.45 αύριο το πρωί για μια σειρά από τις εκθέσεις που θα συζητήσουμε σήμερα. Και να πω ότι αύριο το απόγευμα δεν υπάρχει συνεδρίαση. Να είστε βέβαιοι, να επιβεβαιώσετε μάλλον ότι όντω δεν το έχετε βάλει στι ατζέντε σα. Επίση, αύριο στι 11 και 4 θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Λοιπόν, να περάσουμε στι υπόλοιπε αναγγελίε. Ω συνήθω, να σα θυμίσω ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Να καλωσορίσω λοιπόν το ηλεκτρονικό μας κοινό για σήμερα το απόγευμα και να σας θυμίσω ότι είμαστε πιλωτική επιτροπή για τις συνεδριάσεις άνευ χάρτου. Υπάρχει ηλεκτρονική λοιπόν εκδοχή της συνεδρίασης και των σημειώσεών της διαθέσιμη για όλους τους ε, συναδέλφους, τους βοηθούς και το προσωπικό. Μπορείτε να δείτε δηλαδή όλα τα έγγραφα της συνεδρίασης στο iPad ή στο laptop που έχετε μαζί σας για να γλιτώσουμε όλο αυτό το χαρτί που θα είχατε ιδάλω στα δρανά σα. Εάν θέλετε λοιπόν να, είναι απολύτως, να είστε απολύτω άνευ χάρτου συμμετέχων μέλο τη Επιτροπή, χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή. Να θυμίσω επίση ότι θα γίνει ένα κοκτέιλ για το τέλο τη χρονιά της 6.30 έξω από την αίθουσα συνεδρίαση σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι εκεί. Προφανώς μπορεί να, έρθει και, να έρθουν και οι συνεργάτες μας σε αυτό το κοκτέιλ και έχουμε προσκαλέσει και μια σειρά από επιτρόπους. Ιδίω αυτού με του οποίου συνεργαζόμαστε κατά εξοχήν. Οπότε ελπίζω ότι κάποιοι από του προσκεκλημένου μα θα είναι για αυτό το τελευταίο κοκτέιλ τη χρονιά μαζί μα. Και θα γιορτάσουμε μαζί την επιτυχή εργασία τη Επιτροπή μα. Τη 6.30. Μια ειδική χριστουγεννιάτικη έκδοση του ενημερωτικού μας φυλαδίου του newsletter. Οποιοςδήποτε θέλει να λαμβάνει τακτικά αντίγραφο του, αντίτυπο του newsletter, αρκεί να μας στείλει ένα email μέσω του ιστοτόπου μας. Βλέπετε ότι και μια χριστουγεννιάτικη κάρτα με ένα μήνυμα με ευχές στο πίσω μέρος, οπότε σας το επισημαίνω και αυτό. Τώρα, τα πρακτικά της συνεδριάσεων του Νοεμβρίου. Οι συνάδελφοι τα έχουν στους φακέλους τους και Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει ως προς αυτά, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι είναι εγκεκριμένα. Πριν προχωρήσουμε στην έκθεση της κυρίας Κόλιν ε, Λάγκεν, η πρώτη τη νομοθετική μα για σήμερα το απόγευμα, να σα ενημερώσω για τις διαπραγματεύσει ή να καλέσω του συναδέλφου να μα ενημερώσουν καλύτερα για του τρεμερού διαλόγου. Βλέπω ότι είναι εδώ η κυρία Σάλτε Μόζε. Η κυρία Πιτικάνιαν και εσείς συνεργάζεστε για το θέμα της, ε, της εποπτείας της αγοράς και της ασφάλειας των προϊόντων. Κύριε Σαντεμόζε, αν θέλετε να πάρετε το λόγο για να ενημερώσετε την Επιτροπή για τις προοπτικές του θέματος αυτού και για το πού βρισκόμαστε και πώς μπορεί να προχωρήσει το όλο θέμα. Να υπενθυμίσω ότι μόλις αναθέσαμε στους, ε, μάλλον αναθέσαμε πριν από λίγο καιρό στους συζητητέ μας να διαπραγματευτούν το θέμα αυτό θα ήθελα λοιπόν, επειδή δεν ήμουν πάντοτε εκεί, να μου πείτε τι έγινε σε αυτές τις πραγματεύσει, κύριε Φελντεμόζε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν πραγματικές εξέλιξεις από την τελευταία φορά που είχα έρθει στην Επιτροπή για να το ε, συζητήσω το θέμα αυτό. Έχουμε ακόμη κάποια προβλήματα, όχι από την πλευρά του Κοινοβουλίου, αλλά του Συμβουλίου. Δεν έχουν ακόμη προετοιμάσει πλήρω την εντολή του. Έχουμε συνομιλίε και με τη Λιθουανική Προεδρία και επιδιώκουμε επαφέ και με την ελληνική προεδρία. Θα τους συναντήσω αύριο κιόλα για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, δυνατότητες για διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει πολύ σύντομα να σκεφτούμε ένα χρονοδιάγραμμα για να έρθει στην ε, Ολομέλεια η έκθεση, να ψηφίσει δηλαδή τουλάχιστον η Ολομέλεια. Ακόμη δεν τα έχω παρατήσει, δεν έχω παραδώσει τα όπλα, αλλά Νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πότε θα φτάσει στην ολομέλη έκθεση. Όμω είμαστε διαθέσιμοι ώστε να υπάρξουν διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο εφόσον είναι σε θέση να διαπραγματευτούν και εφόσον λάβουν τέλο πάντων εντολή για τι διαπραγματεύσει αυτέ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κινηθούμε παράλληλα σε δύο οδού για να βεβαιωθούμε ότι δεν χάνουμε την ευκαιρία η έκθεση να ψηφιστεί την Ολομέλεια σε περίπτωση που δεν πετύχουν οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Να πω πάντως ότι το βρίσκω κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί έχουμε εδώ ένα σημαντικότατο νομοθέτημα που θα μπορούσε να αποδώσει ωφέλη και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις και το να μην υπάρξει τελικά συμφωνία απλώς θα μας οδηγήσει σε στο να μην υπάρξει αίσιο πέρα στην εξέλιξη αυτή τη νομοθετική διαδικασία. Και επειδή υπάρχουν και, υπάρχει και επίκενται και ευρωεκλογέ, καλό θα ήταν οι πολίτε να δουν ότι κάτι κάνουμε εδώ. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώ αποφασίζει το Συμβούλιο. Εκείνοι πρέπει να το πάρουν απόφαση αν θα προχωρήσουν ή όχι σε αυτή τη φάση. Του πιέζουμε και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε κάποια απάντηση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πρόεδρος. Ως προς τα προβλήματα θα ήταν ορθό να πει κανεί ότι το θέμα των σημάτων ε, προέλευση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Επιτάπητο, πώς το βλέπετε. Κοιτάξτε, πάνω από όλα είναι το άρθρο 7 με το made in το θέμα, αλλά και κάποιες ε, λεπτομέρειες για την εποπτεία της αγοράς και το σχετικό κανονισμό. Εκεί υπάρχουν όλε τι τριβέ. Αλλά το μέγιστο πρόβλημα είναι ακριβώ το made in. Έχει ακουστεί ήδη εδώ στην Επιτροπή μας και ότι η εντολή μας είναι σαφής, το έχουν πει όλοι, έχουμε συμφωνήσει και με τις σκιώδεις εισηγητές, αλλά παρόλο που θέλουμε τις διαπραγματεύσεις και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, δεν μπορεί να γίνουν διαπραγματεύσεις αν δεν ξεκινήσουν αυτές οι ίδιες. Δεν μπορούμε λοιπόν να προδικάσουμε το τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις πριν περάσουμε σε διαπραγματεύσεις. Απλώ έχουμε δηλώσει την προθυμία μα να διαπραγματευτούμε και ενημέρωσα σήμερα και την Προεδρία. Βεβαίω είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε και για το άρθρο 7, αλλά μέχρι να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι να διαπραγματεύσουν και να αρχίσουν επισήμω διαπραγματεύσει, δεν μπορούμε να πούμε ποιε θα είναι οι παραχωρήσει που μπορούμε να κάνουμε. Σα ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σα και τη συμμερίζομαι. Διότι εσεί και οι υπόλοιποι συγκεκριτέ τη Επιτροπή μα έχετε εργαστεί πολύ σκληρά για να έχουμε γέρο ψηφοφορία στην Επιτροπή και να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει. Και τελικά αυτέ οι διαπραγματεύσει δεν γίνονται. Διότι το Συμβούλιο δεν θέλει να προχωρήσει το θέμα γρήγορα μέχρι το τέλο τη δική μα θητεία. Πάντω, καλώ μα λέτε ότι όντω πρέπει να πιέσουμε μπα και προχωρήσει το θέμα. Δεύτερο του ΣΧΕ, όπου βρίσκονται υπό εξέλιξη διαπραγματεύσει, είναι το θέμα του ραδιοφωνικού εξοπλισμού. Με εισηγήτρια την κυρία Βάιλερ. Δεν είναι εδώ. Απλώς επειδή εγώ προείδρευσα στην τελευταία συνάντηση να σας πω τι έγινε. Είχαμε επικοδομητική συζήτηση όπου επικεντρωθήκαμε στις διαφορές ε, μεταξύ της δικής μας θέσης και αυτής του Συμβουλίου. Τέσσερα βασικά προβλήματα υπήρχαν. Τομείς για τους οποίους προτείναμε λύσει στο Συμβούλιο. Συνάντηση προβλέπεται στις 5 προβλεπόταν στις 5 Δεκεμβρίου, αλλά το Συμβούλιο δεν ήταν έτοιμο ε, για να συνομιλήσουμε και μας ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα μόλις ότι μπορούν να συνεχίσουν τις δημοκρατήσεις. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι μπορεί να επιτελεστεί κάποια πρόοδος. Τελευταίος γύρος τριμερούς διαλόγου με τη Λιβανική Προεδρία λοιπόν θα γίνει την 5η το πρωί στις 18 Δεκεμβρίου και ελπίζουμε ότι η κυρία Βάιλερ θα πάρει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο εκεί. Θα δούμε όμως ε, τι θα γίνει και με το θέμα αυτό. Τώρα έχουμε και την νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις ε, δημόσιες Η κυρία ε, Μπρίκετ Λάγκεν είναι η συγγήτρια, Κόλλιν Λάγκεν, συγγνώμη. Ε, θα ψηφίσουμε για το θέμα αυτό αύριο. Ήδη είχαμε ε, μακροσκελή συζήτηση στην Επιτροπή για το θέμα αυτό και σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε τι συμβαστικέ σα προτάσει. Νομίζω όλε και όλε οι συζητητέ είναι εδώ, εκτό από τον κύριο Κρόιτσμαν, τον κύριο Σταραμπέλα, η κυρία Ρόιλε και εγώ είμαστε εδώ. Δεν ξέρω ποιο θέλει να τοποθετηθεί, όμω και ο κύριο Ροσφόρ από του φιλελεύθερου, βλέπω την εδώ. Αυτό λοιπόν που θα κάνω είναι να δώσω το λόγο στην κυρία Κολυλάνιν για να συζητήσουμε τι τροπολογίε και τι συμβαστικέ τροπολογίε, και μετά θα ακούσουμε και του κέντρου συζητητές για να ε, συζητήσουμε όλοι μαζί. Κυρία Κολυλάνιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την μεγάλη ευρωπαϊκή ηλεκτρονική αγορά, πράγμα το οποίο χαιρετίζουμε. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε προδιαγραφές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Και αυτό θα γίνει εάν συμφωνήσουν όλοι και δεν θελήσουν κάποιοι να απορρίψουν ε, αυτό το θέμα. Βεβαίως πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο τίθεται σε εθελούσια βάση σε εφαρμογή. Αν κάποιος θέλει να το απορρίψει για ένα χύψη λόγο, μπορεί να το κάνει. Πώς έχουν τα πράγματα προς το παρόν. Το Βέλγιο ήδη έχει ένα τέτοιο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης που λειτουργεί. Άλλες χώρες επεξεργάζονται το όλο σύστημα με διαφορετικούς κανόνες, με διαφορετική βάση ίσως δεδομένων. Άρα δεν έχουμε διαλειτουργικότητα και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Μια ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα του όλου συστήματος και εναρμόνιση, ώστε να μπορούν να γίνονται οι συναλλαγές σωστά. Όπως ξέρετε στην πρόταση της Επιτροπής υπάρχουν νέα άρθρα για τα οποία τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις Έχουμε, είχαμε και πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, πράγμα που δεν κατέστησε πιο απλή διαδικασία. Εγώ είχα καταθέσει 33 ε, τροπολογίες και οι σκιώδεις εισηγητές άλλες 23. Στην συνάντηση που είχαμε τους σκιώδεις εισηγητές το συζητήσαμε διεξοδικά το θέμα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους διότι πραγματικά η συνεργασία μας ήταν εξαιρετικά επικοδομητική Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μία συμβιβαστική πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα σχόλια που έγιναν. Θα ήθελα κυρίως να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής γεγονός. Για την ε, αγγλική και γερμανική εκδοχή επίσης πρέπει να σας πω ότι έγιναν κάποιες τροπολογίες που αφορούσαν την γλώσσα αλλά και άλλες που ήταν ουσίας και τις λάβαμε υπόψη. Τώρα, συμβαστική μου πρόταση. Ξεκινώ από την υπόθεση ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε αύριο την ψηφοφορία χωρίς πρόβλημα, δεδομένου ότι όλες οι συμβιβαστικές προτάσεις έγιναν αποδεκτές από τους σκιώδεις εισηγητές. Μέχρι την τελευταία στιγμή με την Άλντε επίσης είχαμε συζητήσει το θέμα ε, μιας ε, νέας ε, πρότασης στο 8 δέλτα και πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει και εκεί κανένα πρόβλημα. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω. Τα κείμενα τα οποία σας έχουν διανεμηθεί δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό το 8 β, με συγχωρείτε, όχι δέλτα, δεδομένου ότι η γραμματεία βρισκόταν στην φάση της εκπόνησής του πριν να τυπωθεί. Γι' αυτό Περνάω αμέσως στην ε, εξέταση των ε, συμβιβαστικών προτάσεων. Πρώτα απ' όλα στο άρθρο 3 έχουμε καταρτήσει κατάλογο στον οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν το χρονοδιάγραμμα, το ΣΕΝ, την ε, προθεσμία των 24 μηνών για να μπορέσει να δημιουργηθεί ε, αυτή το ΣΕΝ, το European Standardization Organization. Είπαμε επίσης ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται μεταξύ ε, των επιχειρήσεων που θα πρέπει να κάνουν κατά την διάρκεια 6 μηνών τις ε, δοκιμές μεταξύ τους για να δουν εάν ε, ε, μπορέσουν να έχουν ε, ολοκληρώσει επιτυχώς όλες αυτές τις, το σύνολο των κανόνων, επίσης προβλέπονται τρεις μήνες για να μπορέσει η Επιτροπή να εκπονήσει την πρότασή της και από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή πιλωτικά η, η νόρμα αυτή για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέχρι την, το τέλος της εφαρμογής θα, υπάρχουν, υπάρχει χρονική διάρκεια 63 μηνών. Ε, Επίσης, κατά τη διάρκεια των δοκιμών που θα γίνουν, θα πρέπει, όπως ε, λέγεται, να υπάρχει ε, ευκολία στην εφαρμογή της. Προβλέπεται επίσης ε, χρόνος για να μπορέσει να μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια η εφαρμογή αυτής της της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ήδη έχουν ε, κατά κάποιο τρόπο ε, θέσει σε εφαρμογή αυτά τα πρότυπα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται λοιπόν στην πρόταση, στις διάφορες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί κυρίως οι προβλεπόμενες προθεσμίες που πήγαιναν από 18 έως 36 μήνες και εδώ υπάρχουν διάφορες διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Εγώ είχα προβλέψει 15 μήνες για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και 15 συμπληρωματικούς για τις διάφορες μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές. Γι' αυτό είχα καταρχάς Ε, φτάσει στο τέλος λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαδικασίες σε 66 ε, μήνες. Εν πάση περιπτώσει όμως η Κομισιό είναι αυτή η οποία θα πρέπει να κάνει τον όλο φάκελο να προχωρήσει. Αυτά ήθελα να πω πρόεδρε αρχίζοντας. Σας ευχαριστώ για τις σαφείς σας ε, εξηγήσεις και για τις συμβιβαστικές τροπολογίες που συμπεριλάβατε στην, στην πρόταση συμβιβασμού. Ο κύριος Στάμπα επίσης είναι εδώ από την ε, Κομισιό. Τον καλωσορίζω και όταν θα του δώσω το λόγο για να κάνει τις διά, τα διάφορα σχόλια όσον αφορά τις βασικές τροπολογίες. Ο κύριος Ταραμπέλα, ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση εμπλουτίζει διευκολύνει την ηλεκτρονική αγορά στον τομέα συγκεκριμένα των δημοσίων συμβάσεων. Όπως ξέρουμε, το θέμα αυτό θα συζητηθεί το απόγευμα της 14ης Ιανουαρίας στην Ολομέλη και θα ψηφιστεί στις 15. Περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό Έγινε στην ΙΜΚΟ πρώτη ψηφοφορία της 5 Σεπτεμβρίου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στο τέλος με, να ολοκληρώσουμε τη δικασία με επιτυχία και να πιούμε και ένα ποτηράκι. Τώρα, για τις δημόσιες συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τι έχει γίνει στα δύο κείμενα αυτά, ώστε να μπορέσουν να έχουμε ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, θα πω ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις από αυτή την εφαρμογή στην δημόσια δίκαιση κυρίως για την διαφάνεια των διαδικαστικών, για την μείωση του κόστους και αυτά είναι πλεονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίσουν όλοι οι οικονομικά εμπλεκόμενοι. Εκ μέρους της S&D ως κοιόδης συζητητής εγώ είχα ε, προτείνει Διάφορε τροπολογίε για να διευκολυνθούμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίηση. Είχα μιλήσει για μειωμένη προθεσμία εφαρμογή, εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, ώστε να μην υπάρχει συμπληρωματικό κόστος για τους δικαιούχους αυτή τη οδηγία. Τώρα, ελήφθη υπόψη, όπω είπε η κυρία Λάγκεν, οι διάφορες προτάσεις που έκαναν οι συνάδελφοι, εν μέρη τουλάχιστον, δεδομένου ότι πρόκειται για συμβιβαστική πρόταση, πρέπει να πω ότι παρόλα αυτά οι προθεσμίες ε, μειώθηκαν, αλλά και παρόλα αυτά εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ εκτενείς και για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για, τους μη, για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές. Ε, και βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για ε, μεγαλύτερη απλοποίηση της όλης διαδικασίας στη διάρκεια κυρίως μεταβατικής περίοδου. Η φάση επίσης του τεστ της δοκιμής είναι πολύ σημαντική. Μας έπεισε με τα επιχειρήματά της η εισηγήτρια. Ε, Επίση, όπως είπε ο κύριος Κρότσμαν και εγώ, θα πρέπει στο σημείο 8 να ε, έχουμε μια καλύτερη διατύπωση, πιο σαφή και θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο διότι με μεγάλη ταχύτητα και απόλυτη σαφήνεια μετέφερε όλες τις ιδέες. Γι' αυτό θα ήθελα ευχαριστώντας σας να σας πω ότι δέχομαι την ε, συμβιβαστική πρόταση που κάνετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι. Και εμεί αναμένουμε την ψηφοφορία για το, για το σύνολο του πακέτου. Όπως είπατε, θα γίνει στην ε, Ολομέλεια του Ιανουαρίου η συζήτηση, τρίτη η ψηφοφορία την Τετάρτη. 14 και 15 Ιανουαρίου θα δείτε στη μερίδα διάταξη όλες τις λεπτομέρειες. Όλοι όσοι λοιπόν ε, ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των δημοσίων συμβάσεων, θα βρουν τα σχετικά στοιχεία στο ίντερνετ. Και είδατε ότι το κάνουμε στην καλύτερη δυνατή ώρα, στην ώρα μεγάλου ενδιαφέροντος, στην συζήτηση και την ψηφοφορία. Ο κύριος Γοξφό ε, αντί του κύριου Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Κρόιτσμαν που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα το απόγευμα. Μου ανέθεσε να σας παρουσιάσω τις παρατήσεις του. Θα ήθελε προφανώς να ευχαριστήσει την εισηγήτρια καθώς και τους κοιόδες εισηγητές για την εργασία που επιτέλωσαν και την επικοδομητική συνεργασία όπως υπογράμμισε και ο Μάρκ Ταραμπέλα προηγουμένως μεταξύ όλων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ποια ήταν η φιλοσοφία που άπτεται των προτάσεων που έκανε εξ ονόματος της Άλτε. Με τις τροπολογίες του κύριος Κρόιτσμαν θέλησε αυτό το νέο πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης να εγγυάται την προστασία δεδομένων κυρίως των προσωπικών και να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και τις ανάγκες όλων των αναθεσουσών αρχών που είναι πολυάριθμες με ε, διαφορετικό ε, καθεστώς και διαφορετικές όσον αφορά την διάστασή τους. Θα πρέπει να μπορούν ε, σε, στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στο B2B επίσης να εφαρμόζονται αυτού του διαδικασίες, να είναι συμπληρωματικές και να είναι και συμβατές με, τις, με τα διεθνή πρότυπα επί του θέματος αυτού. Χαιρετίζει το γεγονό ότι όπω είπατε και προηγουμένω η εισηγήτρια συμπεριέλαβε τι προτάσει του στην συμβαστική πρόταση την οποία υποβάλλει. Βεβαίω, όσον αφορά την ε, μεταφορά σε κάθε εθνικό δίκαιο που είναι κάτι το οποίο συζητούμε εδώ, ο συνάδελφος τονίζει Όπω είπε και η συγγήτρια, για τις προθεσμίες να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των αναθετουσών αρχών, κυρίως των μικρών. Αλλά είπε ότι το κόστος θα πρέπει για όλους να είναι περιορισμένο και ε, εάν μπορούμε, οι προθεσμίες αυτές, ε, αν μπορούμε τις προθεσμίες αυτές να τις ε, περιορίσουμε σε λιγότερες μήνες, να το κάνουμε. Η τελευταία συμβιβαστική λύση που αναφέρατε, το 15 συν 15 μήνες, δεν ε, ανταποκρίνεται στην αρχική ιδέα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλύτερη στην πρώτη πρόταση της εισηγήτρια, 18 συν 18 μήνες. Μας φαίνεται λοιπόν ότι είναι το 15 συν 15 αποδεκτό. Επίσης χαιρετίζει την ε, ε, δική σας πρόταση ώστε να μειωθεί και η προθεσμία, τη μεταβατική περίοδος 24 μήνες αντί των 30 που προβλέπονταν στην αρχή και να αποσαφινίστηκε στην έκθεση διάφορες αιτιολογικές σκέψεις ώστε κατά διάρκεια της Διαδικασία μεταφορά σε κάθε εθνικό δίκαιο να είναι τα πάντα σαφή ώστε να μην χαθεί περαιτέρω χρόνος. Σας ευχαριστώ. Η Άλτε, όπως καταλαβαίνετε, υποστορίζει όλες τις συμβαστικέ τροπολογίες που κατατέθηκαν από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και ευχαριστώ την κυρία Λίγκεν για την υπομονή της και για το ότι υποστήριξε το φακελό της. Νομίζω ότι τώρα δεν θα υπάρξει άλλη συνεδρίαση. Νομίζω ότι αυτή η φάση δοκιμής είναι εξαιρετικά σημαντική και θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Αν λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει πρόσθετο κόστος, αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει ε, να τηρήσουμε τις λογικές προθεσμίες, να μην είναι οι προθεσμίες πολύ μικρές, διότι αυτό θα αυξήσει το κόστος. Νομίζω ότι ο συμβιβασμός θα παραμείνει ως έχει άθικτος. Εγώ είμαι ε, για προθεσμίες που θα είναι μεγαλύτερες. Ευχαριστώ πολύ. Για να συμπληρώσουμε με τους σκιώδεις, είμαι και εγώ σκιώδης, θα ήθελα να επιβεβαιώσω και εγώ ότι συμφωνώ με το όσα λέχθηκαν από την κυρία Λάγκεν ε, και εργάστηκε σκληρά για να ενσωματώσει σημαντικές ε, ιδέες που ενδυναμώνουν αυτήν την πρόταση και υποστηρίζουμε την όλη προσέγγιση για την δοκιμή. Άλλες απόψεις που ήταν σημαντικές τώρα έχουν περιληφθεί στο συμβιβασμό ε, σχετικά με την συνεκτικότητα με όλη την χρήση από τη μια άκρη στην άλλη ε, της ηλεκτρονικής ε, τομολόγησης Τιμολόγηση για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά και για μετέπειτα συναλλαγές, διότι η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι σημαντική. Δεν είναι μόνο για την φάση των συμβάσεων, αλλά έχουμε μετά τις, τα τιμολόγια, τις πληρωμές που εμπεριέχουν ε, πάρα πολλές συναλλαγές, δραστηριότητες συναλλαγών. Ε, δεν ε, είναι μόνο ε, για τις δημόσιες συμβάσεις και την αρχική ανάθεση το θέμα αυτό. Θα πρέπει το όλο κόστος λειτουργίας των συμβάσεων να είναι πιο αποτελεσματικό, γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης η οδηγία θα απαιτήσει οι δημόσιες αρχές να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τα τιμολόγια με το σύστημα αυτό το ηλεκτρονικό. Κάναμε λοιπόν μερικές αλλαγές και κάναμε μερικές ειδικέ ε, προτάσεις ε, σχετικά με τα συμβόλαια. Η κυρία Λάγκεν και οι σκιώδεις εισηγητές ε, τις δεχτήκαν αυτές. Θα το δούμε αύριο τι θα γίνει με την ψηφοφορία. Πρωτού δώσω τον λόγο στην Επιτροπή. Θέλει κανένα άλλος συνάδελφος να σχολιάσει. Θα καλέσω τον κύριο Στάμπερντ να πει μερικά λόγια εξ ονόματος της Κομισιόν, να μας πει τι σκέφτεται για την εργασία μας σχετικά με το θέμα αυτό και του συμβιβασμού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και κυρίως την κυρία Κολίν Λάγκαν και τους σκιώδεις εισηγητές για την σημαντική εργασία την οποία επετέλεσαν. Κυρίως με, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ούτως ώστε να αποπερατώσουμε αυτές τις προτάσεις ε, και η ταχύτητα της εργασίας του Κοινοβουλίου είναι ευπρόσδεκτη. Πιστεύουμε επίσης ότι η πρόταση βελτιώθηκε από πολλές απόψεις και χαιρετίζουμε ιδιαίτερα αυτό που λέχθηκε για την προστασία των δεδομένων είναι κάτι σημαντικό επίσης για τις δοκιμές. Το θέμα αυτό που προτάθηκε από την εισηγήτρια είναι νομίζουμε ένα θετικό στοιχείο για την όλη διαδικασία. Είναι σημαντικό αυτό που σχεδιάζεται και αυτό που θα προκύψει από την τυποποίηση να είναι κάτι το χρήσιμο για τις συμβαλόμενες αρχές. Βεβαίως από την αρχή όσον αφορά τη δοκιμή θέλαμε να αποφύγουμε, να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις και στην διαδικασία τυποποίησης περιλαμβάνεται το στάδιο της δοκιμής και αυτό είναι ένα βήμα θετικό. Έχουμε ακόμα ορισμένα πράγματα που θα πρέπει να διευκρινιστούν ως προς τη δοκιμή στον τρίμερη διάλογο. Υπάρχει κάποια παρεξήγηση ε, για το τι θα πρέπει να δοκιμάσουμε, να θέσουμε υποδοκιμή. Είναι τα πρότυπα, είναι όμως κάτι το τεχνικό που θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε στο επίπεδο του τριμερούς διαλόγου. Αλλά πάντως ε, είναι ε, μια συνεισφορά θετική. Σημειώσαμε και συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό για την ανάγκη οι συνομοθέτες να έχουν μια καλύτερη συμμετοχή, όχι αφού υπογραφεί η οδηγία και υιοθετηθεί, αλλά πριν. Σε κάποιο στάδιο αφού θα έχουν αναπτυχθεί τα πρότυπα ή τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το σημειώνουμε αυτό. Δεχόμαστε καταρχήν την ιδέα και πιστεύουμε ότι το άρθρο 11 της νομοθεσίας περί τυποποίησης είναι ένας κατάλληλος μηχανισμός που το εξασφαλίζει αυτό ε, και πιο γενικά και αυτό θα συζητηθεί στον τριμερή διάλογο και αυτό είναι σημαντικό για μας είναι αυτή η συμμετοχή και ο έλεγχος των συνομοθετών να παραμείνει στο πλαίσιο των όσων έχουν γίνει ε, δεκτά στα πλαίσια της νομοθεσίας περί τυποποίησης. Βεβαίω, αυτό θα το διερευνήσουμε, θα το μελετήσουμε περαιτέρω στον τριμερή διάλογο. Ο τομέα όπου έχουμε κάποιε ανησυχίε, και αυτό θα αποτελέσει στο αντικείμενο ε, δυσκόλων ε, διαπραγματεύσεων είναι ο χρονισμός, τα χρονικά περιθώρια. Πρέπει νομίζουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν μικρότερες τις προθεσμίες. Κατανοούμε βεβαίως ότι οι συμβαλόμενες αρχές, περιφερειακές, τοπικές, ίσως χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Λαμβάνουμε υπόψη το σημείο αυτό, αλλά ο χρονισμός που έχουμε τώρα επιτάπητος είναι αρκετά μεγάλος, μας οδηγεί μακριά και ένα από τα πράγματα τα οποία μας ενοχλεί είναι ότι ε, δεν ε, συμμορφωνόμαστε τώρα με τις δεσμεύσεις του πακέτου δημοσίων συμβάσεων και επειδή αυτό βρίσκεται σε τεχνικό επίπεδο με όλες τις ηλεκτρονικές φάσεις ε, ανάθεση, συμβάσεις κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει καμιά εναρμόνιση ανάμεσα σε αυτό που συμφωνούμε εδώ για την τιμολόγηση. Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη επειδή όλοι είμαστε πεπισμένοι για την σημασία αυτού του νομοθετήματος ε, που πρέπει να συμπληρώσουμε ε, τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και όλοι το επιθυμούν αυτό γύρω από το τραπέζι, και όλοι επιθυμούν μια συμφωνία και έχουμε την πεποίθηση ότι στον επόμενο τριμερή διάλογο θα το επιτύχουμε αυτό. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την θετική σας ανταπόκριση. Περιμένετε βεβαίως έναν τριμερή διάλογο. Θα πρέπει βεβαίως τυπικά να λάβουμε αυτή την απόφαση που εξαρτάται και από την και όλη κυρία Κόλιν Λάγκεν και τους σκιώδεις συζητητές. Η κυρία Κόλλιν Λάγκεν θα μπορούσε να συνοψίσει και να μας πει ποια είναι η στρατηγική της όσον αφορά στο Συμβούλιο και αν ε, έχει συζήτηση με την ελληνική Προεδρία ε, και ποια είναι η εικόνα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπαν οι σκιώδεις εισηγητές ε, είναι επικαλυπτόμεθα όλοι, δεν έχω ιδιαίτερο σχόλιο, όλοι συμφωνούμε, δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την ελληνική προεδρία. Ήθελα πρώτα απ' όλα ε, να συμμετάσχω σε αυτή την συνεδρίαση. Ε, θα μπορούμε, μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη στρατηγική, αλλά το βασικό σημείο θα είναι ότι η προθεσμίας θα πρέπει να διευκρινιστούν για την υλοποίηση. Άλλη μια ερώτηση που θα θέλω να θέσω στην Κομισιό βρίσκω ότι αυτό που είπε ο κύριος Ταραμπέλα με εκπλήσει κάπως, το είχε ήδη προτείνει, είπατε κύριε Ταραμπέλα ότι θα έπρεπε να καταστεί δυνατόν για τα πρότυπα να έχουμε μια διαδικασία που θα μπορούν να την διαχειριστούν καλύτερα οι τοπικές αρχές, αλλά διαρωτώ αυτό το πράγμα είναι εφαρμόσιμο, μπορούμε να το διανοηθούμε και αν ναι θα ήθελα να έχουμε μια απλουστευμένη διαδικασία με το σύστημα αυτό. Πολύ καλά. Θέλετε μια απάντηση από την Κομισιό. Well, Και πάλι και αυτό αποτελεί μέρος της τεχνικής συζήτησης που θα έχουμε. Αν καταλαβαίνετε το πρότυπο ε, με το λιγότερο περιεχόμενο δεν ε, βλέπω να το έχουμε αυτό με τον ένα ή άλλο τρόπο. Έχετε και τη τη σύνταξη και την χαρτογράφηση εκτός από το πρότυπο που ε, προβλέπει πόσο το περιεχόμενο αυτό θα ενταχθεί με ηλεκτρονική γλώσσα. Και νομίζω ότι αυτά τα διάφορα προγράμματα, οι διάφορες συντάξεις συντακτικά ε, που θα, ε, που θα εντάξουν το, όλα το πρότυπο θα μπορούν ε, να φορτωθούν. Δεν βλέπω καμία τεχνική δυσκολία. Δεν ξέρω αν αυτό θα καταστήσει τα πράγματα ευκολότερα. Εκεί έγκυται νομίζω η δυσκολία κατά τη γνώμη μου. Αλλά ίσως μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά διμερώς. Πολύ καλά. θα συναντήσουμε, συναντήσετε ίσως την ελληνική προεδρία και ίσως θα μπορείτε να ζητήσετε από την Επιτροπή μας να σας δώσει μία εντολή για να συνεχιστούν οι συζητήσεις ή αλλιώ αυτό θα πρέπει να γίνει τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ πολύ όσους συμμετείχαν. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε αύριο και μετά υποθέτοντας ότι συμφωνεί η Επιτροπή μας θα, προς, ε, προσφέρουμε να ανοίξουν διαπραγματεύσεις ε, με ε, το Συμβούλιο. μήπως να μπορούμε να έχουμε συμφωνία πριν από την αρχή του Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποπερατώσουμε τις εργασίες το Φεβρουάριο, ίσως πριν αν θέλετε τις, τις εκλογές και θα είναι το, η έκθεσή σας κυρία Κόλιν Λάγκεν που θα έχει αυτό το προνόμιο. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Μια έκθεση από την Επιτροπή μας αποκρισή στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, τυποποίηση, για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας, ο κύριος Ροσφόρη είναι ο εισηγητής. Και έχουμε σχεδόν αρκετέ στην κυρία Σινέλοβα που δεν τη βλέπω, την κυρία Ρόιλε όμω είναι εδώ, εγώ είμαι εδώ, ο κύριο Μπόρισοφ. Οπότε Α προχωρήσουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετέ συμβαστικέ τροπολογίε. Θα ήταν καλό η να τι παρουσιάσει. Υπάρχει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε φαντάζομαι ότι και εσείς τα σχολιάσετε τι συμβαστικέ τροπολογίε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ροσφόρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, η έκθεση αυτή είναι σημαντική. Την έχουμε συζητήσει επανειλημμένως στην Επιτροπή μας. Είχαμε 60 τροπολογίες προς εξέταση, 14 που τις είχα υποβάλει εγώ ως εισηγητής. Και ναι, είμαστε ικανοποιημένοι που καταλήξαμε σε 8 συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες θα ψηφιστούν αύριο το πρωί από την Επιτροπή μας. Οι συμβαστικέ αυτέ τροπολογίε στηρίζονται από την πλειονότητα των συναδέλφων. Του ευχαριστώ λοιπόν θερμά για την καλή μα συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία. Εάν μου επιτρέπετε, θα σταθώ στα σημαντικότερα στοιχεία των συμβαστικών τροπολογιών. Η πρώτη τροπολογία είναι συντακτική υφή, οπότε την αφήνω κατά μέρο. Η συμβαστική δύο αφορά το θέμα των ε, προσωρινών παρεκκλήσεων για την, υλοποίηση, για την εφαρμογή της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν θεωρεί απαραίτητο να επανέλθουμε στο σημείο αυτό. Συμφωνούμε μαζί τη, αλλά ζητούμε ρητό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει νέα έκθεση εφαρμογή σε μία διετία ιδιαίτερο για να βεβαιωθούμε ότι η οδηγία όχι απλώ ε, εφαρμόζεται σωστά, αλλά επιτρέπει να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο ε, προστασία των καταναλωτών. Γιατί θα θυμάστε ένα από τα μέγιστα προβλήματα στην εφαρμογή τη οδηγία αυτή ήταν ακριβώ το θέμα τη υλοποίησή τη και όχι τόσο το θέμα του πλαισίου ε, εντό του οποίου καθορίζει τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Μια από τις βασικές μας μέρημνες μεταξύ των συναδέλφων του ΕΛΚ ήταν η έκθεση αυτή να αξιολογήσει και την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνιση κατά την εφαρμογή τη οδηγία αυτή. Νομίζω ότι στο σχετικό εδάφιο προσπαθήσαμε να, ε, και ελπίζω το πετύχουμε, προσπαθήσαμε λοιπόν να καθησυχάσουμε αυτέ τι ανησυχίε. Οι συμβαστικέ 3 και 4 αφορούν το θέμα τη συνεργασία μεταξύ των ε, των εθνικών αρχών θα δείτε ότι και αυτό είναι ζωτικής σημασίας σήμερα, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες, απλώς να θυμίσω, να διευκρινίσω μάλλον, ότι σε ό,τι αφορά τη συμβαστική 4, υπάρχει μια ιδέα να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ε, επιμέρους κρατών με μια επιπλέον μία στις ε, τρέχουσες διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού ε, συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών. Θυμίζει όλα τα, όλες τις συμμετέχοντες πλευρές που ενεργώς θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις συνομιλίες, τις διαβουλεύσεις. Η συμβαστική 5 αφορά το θέμα των κυρώσεων Προφανώς για να είναι αποτελεσματική η εργασία μας όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπάρχουν αποτρεπτικές κυρώσεις. Και σήμερα δεν είναι πολύ σε αυτά τα πράγματα ω προς τις κυρώσεις. Γι' αυτό ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να εξετάζει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν για τις κυρώσεις που ισχύουν και το πώς εφαρμόζονται, πώς επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη. Εδώ νομίζω και η τροπολογία αυτή είναι ικανοποιητική γιατί στην διατύπωσή της υπάρχει κάλυψη των διαφορετικών προτεραιοτήτων των ε, μεν και των δε. Η έκτη συμβαστική τροπολογία αφορά τα ε, έγγραφα προς ανατολισμό, ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν πολλές καλές ιδέες που έχουν διατυπωθεί από τους συναδέλφους και συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις συμβαστικές. Ιδιαίτερως θυμίζω την ε, συστηματική επικαιροποίηση των εγγράφων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια διαδικασία μεγάλης διαφάνειας και την ε, ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εθνικών αρχών. Η συμβαστική 7 αφορά ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο. Το θέμα της εμπορικής προώθησης και των σχετικών πωλήσεων. Ή μάλλον των ε, συνδεόμενων πωλήσεων. Εδώ θυμάστε ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν αυτομάτως παράνομες, ούτε περιλαμβάνονται στο πρώτο παράρτημα που ε, ανακεφαλαιώνει συνοψίζει τι απαγορευμένε πρακτικέ. Από πολλά κράτη-μέλη όμω, όπω το δικό μου, δεν μπορεί να υπάρξει αυτή καθεαυτή η απαγόρευση. Υπάρχει μεγάλο επίπεδο, πολύ ψηλό επίπεδο επίβλεψη για να εμποδίζονται αυτέ τι εμπορικέ πρακτικέ. και εδώ ζητάτε να υπάρξει ε, αναπερίπτωση αξιολόγηση για να δούμε πότε ακριβώς αυτές οι πρακτικές μπορεί να είναι παραλαπλανητικές ή επιθετικές. Εάν δεν συμβαίνει αυτό και αν αντίκειται στους κανόνες του επαγγελματικού, ε, της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας θα πρέπει να επιτρέπονται για να μην ε, παρεμποδίζεται και η δυνατότητα του καταναλωτή να παρακολουθεί την οικονομική του ακαιρεότητα. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει υπό ποιου όρου αυτέ οι πρακτικέ γίνονται παράνομες με το πλέον κατάλληλο εργαλείο, αυτό που θα θεωρήσει εκείνη απαραίτητο, το οποίο θα μπορούσε να συμπεριλάβει σε ένα έγγραφο προσανατολισμού ή να ε, συλλάβει μια άλλη ιδέα για ένα νέο ενδεχομένω νομοθετικό εργαλείο που να καλύπτει ακριβώ αυτή την ανάγκη. Η συμβιβαστική υπαριθμών 8 αφορά το θέμα των συλλογικών προσφυγών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερω που επί τη τροπολογία αυτή υπήρξε μεγάλη στήριξη Τώρα αν δεν συμφωνούν απολύτω όλε οι, οι πολιτικές ομάδες, αυτό είναι άλλο, αλλά γενικώ υπάρχει μεγάλη συμφωνία στα πλαίσια μιας, ε, μιας γενικής συζήτησης για τι ομαδικές προσφυγέ, και καταφέραμε βαθμιδό να περάσουμε στην υλοποίηση και ενό τέτοιου εργαλείου και ελπίζουμε θα πετύχει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οκτώ λοιπόν συμβαστικέ τροπολογίε, ολοκληρώνοντα. Να θυμίσω ένα άλλο θέμα που επίσης το συζητήσαμε διαμακρών στην Επιτροπή μας, το πώς όλα αυτά θα επεκταθούν και στις επιχειρήσεις, στο B2B. Εδώ δεν ε, υπέβαλα συμβαστική τροπολογία, όμως είμαι θετικά διακείμενος προς τις ε, τροπολογίες του κ. Χάρμπορ, της κ. Ε, Γκρίπ και νομίζω ότι θα μπορέσω να τις στηρίξω. Όπω το είπα πανελειμμένω, δεν ήμουν ευνοϊκό προ την ε, πρόταση του κ. Νταγιούν το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία να να διευρυνθεί και στον τομέα B2B. Για τους λόγους που είχα προαναφέρει. Τα κράτη-μέλη, εάν το επιθυμούσαν, μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρή ζήτηση ώστε η δυνατότητα αυτή να προβλεφθεί και να γενικευθεί. Εδώ, Πρόεδρε, συνοψίζοντας τι καταφέραμε να πετύχουμε, νομίζω ότι ήταν ποιοτική η εργασία μας και περιμένω να ακούσω και τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών συναδέλφων, καθώς και των υπολείπων συναδέλφων που θέλουν ενδεχομένω να τοποθετηθούν για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ ξανά όλους για την εξαιρετική μας συνεργασία. Θα τα ξαναπούμε προφανώς αύριο για να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή, αλλά νομίζω και στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου, όλα πάνε καλά, για την έγκριση, την τελική έγκριση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε για την ε, διεξοδική αυτή παρουσίαση. Είστε πολύ κατάλληλο άνθρωπο να μιλάτε για τα θέματα αυτά, διότι είστε και ο πλέον ειδικό. Κύριε Μπόρισοφ, πρόεδρε, κύριε Ρώσφου, κατά πρώτον να σα ευχαριστήσω για την πολύ καλή καρποφόρα εργασία που είχαμε. Δεν, έχουμε πολλές, δεν πολλέ αντιρρήσει από την πλευρά του ΕΛΚ για την πλήρη αναδμόνηση θα συμφωνήσω με τη συμβαστική τροπολογία 2 που καλεί τα κατημέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία στα δυνατόν συντομότερα. Επίση, θα συμφωνήσω με τη νέα εκδοχή τη τροπολογία, η οποία αρχικά μα δημιουργούσε προβλήματα. Μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση των σοσιαλιστών και δημοκρατών να ζητήσουν το περαιτέρω διευκρίνηση του θέματο αυτού στο παράρτημα 1. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μια νέα έκθεση για την υλοποίηση τη οδηγία σε μια διετία, προκειμένου να διασφαλίσει και να επιβάλλει την σωστή εφαρμογή. Τώρα για την συμβαστική έξι και τα έγγραφο προσανατολισμού. Ε, πρέπει να μα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα έγγραφα αυτά όντω θα είναι χρήσιμα και όντω ε, ζητούμε ω ΕΛΚ να αναθεωρηθεί το σημείο αυτό στο 2014. Θα πρέπει λοιπόν σε συστηματική βάση να ενημερώνονται τα κατημέλη για το πώ προχωράει η εφαρμογή τη οδηγία αυτή. Σε ό,τι αφορά τι συλλογικέ προσφυγέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σφάτ, τον κύριο Ζάκ και τον κύριο Ρόσφορ για την. Ε, εντατική του δουλειά στο θέμα αυτό. Στην συμβαστική αυτή ζητούμε από τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία οργάνων εξέταση των συλλογικών προσφυγών. Εδώ όμω πρέπει να αποτιμήσουμε το κατά πόσο νομοθετική αυτή πρόταση ε, μπορεί να, πρέπει να γίνει ξεχωριστά με ειδικά δικά τη ε, μέσα θα πρέπει να δούμε όλες τις δυνατότητες ε, ομαδικής προσφυγής και το κατά πόσον αυτές προχωρούν σωστά. ώστε να αποφύγουμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει αυστηρότερη εφαρμογή και καλύτερη υλοποίηση, ώστε οι ενώσεις των καταναλωτών να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, αλλά να προστατεύονται ο εμπορικό και ο ε, και οικονομικός τομέας, καθώς επίσης να υπάρχει ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Αυτά. Η ε, κυρία Σανάλοβα δεν είναι εδώ. Η κυρία Σανάλοβα, όχι, είναι εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους υπόλοιπους τους εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε ε, προκειμένου να εξεύρουμε αυτές τις συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την άριστη συνεργασία. Ε, καταφέραμε να ετοιμάσουμε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες σε γενικές γραμμές μπορούμε να αποδεχτούμε υπογραμμίσαμε ότι η μεγαλύτερη απέτηση, η πιο σημαντική απέτηση είναι η εφαρμογή ε, του δικαίου και των κανόνων μας ακόμα και στις διασυνοριακές συναλλαγές. Η έννοια συμμετοχή των ενώσεων των καταναλωτών είναι πολύ σημαντικό, συμβαστική πρόταση 3. Συμφωνώ με όλα όσα αφορούν την ε, αξιολόγηση των απαγορευμένων πρακτικών που εντάσσονται ή όχι στις ε, παράνομες, στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, συμβαστική δύο και που θα πρέπει να αξιολογηθούν αναγκάτως μέλος. Συμφωνούμε λοιπόν με αυτή την τροπολογία, αλλά να επιμείνω περαιτέρω άλλες δύο τροπολογίες, την 7 και 60, δικές μου τροπολογίες, για τις οποίες θέλω να ζητήσω από τον συνάδελφο να τις υποστηρίξει. Η έκθεση αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η αφορμή. Εκεί θα πρέπει να αναλυθούν και να μελετηθούν οι επιθετικές πρακτικές. Τα κράτη-μέλη αναφέρουν ότι η επιθετική τακτική συνήθως εφαρμόζεται εκτός καταστημάτων, εκτός εμπορικών ε, καταστημάτων. Θα πρέπει εδώ να δώσει μια ιδιαίτερη προσοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι αυτό θα βελτιώσει τη θέση των ε, εμπόρων που εφαρμόζουν ε, το νόμο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει πρωτομέλημα την προστασία των καταναλωτών. Είναι ένας από αυτούς τους, ο τομέας αυτός είναι ένας από τους πλέον προβληματικούς. Ιδίω ό,τι αφορά την πόλη τροφίμων, αλλά και άλλους τομείς. Είναι ένα απλό παράδειγμα αυτό. Δεν πρόκειται για έναν διεξοδικό διάλογο. Αυτές είναι οι δικές μου τροπολογίες και θα σας παρακολουθήσω να τι υποστηρίξετε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν υπογράψαμε διότι είχαμε και εμείς καταθέσει τροπολογίες, άρα δεν ήταν λογικό. Παρ' όλα αυτά τις υποστηρίζουμε, διότι πιστεύουμε ότι είναι καλές. Και εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι η παρατήρησή σας για το B2B είναι σωστή. Το είχα πει εξάλλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δεν ξέρω αν θα διαθετήσουμε το θέμα αυτό σε αυτή την οδηγία, αλλά εν πάση το επιχείρημά σας είναι σωστό και θα σας υποστηρίξω. Επίσης, χαίρομαι διότι σιγά σιγά καταλήγουμε σε συμβιβαστική λύση όσον αφορά τις συλλογικές δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες που καταβάλατε, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο το όλο θέμα και γι' αυτό και πάλι σας ευχαριστώ. στην ε, τροπολογία 2 γίνεται με ε, σχετική πρόταση για εναρμόνιση και απλούστευση της όλης διαδικασίας. Βεβαίω, εάν πρόκειται για συμπληρωματική νομοθετική πράξη, έχει καλό σε περιπτώσει. Γενικότερα όμως, συμφωνούμε με την ε, άποψη του εισηγητή για, την, για το B2B, την ε, επέκταση του συστήματος στο B2B. Αλλά σε κάποιες από τις τροπολογίες μας που ελπίζουν τα υποστηρίξει ο θέλουμε να ενισχυθεί ε, η δράση της Επιτροπής για την αθέμητη πρόθεση και διαφήμιση που ακολουθείται. Και κυρίως αυτές που εφαρμόζονται όταν κανείς ε, συμβουλεύεται τους ε, καταλόγους που έχει στη διάθεσή της κάποια επιχείρηση για να κάνει τέτοιο είδους έμεση διαφήμιση ίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το γεγονό ότι θέλουμε να ληφθεί δράση χρησιμοποιώντας τα κοινοτικά μέσα που διαθέτουμε και θα θέλαμε η Επιτροπή να μας το σχολιάσει αυτό το θέμα. Κατά την άποψή μου όμως αύριο θα γίνει σωστή επικοδομητική ψηφοφορία και πιστεύω ότι με τις συμβαστικές τροπολογίες θα επιτύχετε την πολιτική σύμβαση. Κύριε Μπορισό, θέλετε πάλι κάτι να πείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Δεχτήκαμε εμείς το θέμα ε, αυτό των ευρώ πρέπει να γίνουν κυρίως στον τομέα τον οποίο έχει εντοπίσει η Κομισιό. Ε, δεν ξέρω αν ανέφερε κάτι παρεμφερές η σοσιαλιστική ομάδα. Εμείς εδώ θα θέλαμε να περιοριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προηγούμενους ομιλητές. Το θέμα που ανέφερε ο κύριος ε, ε Πρόεδρος για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Θα ήθελα να υποστηρίξω τα που γιατί έχει επιπτώσεις από αυτές τις ε, πολύ ε, κακές ε, εταιρείες που υπάρχουν ε, οι οποίες με υποχθόνιο τρόπο φτάνουν σε εσά και σε λένε κάποια πράγματα υποχρεωτικά πρέπει να τα κάνετε. Θα ήθελα κάτι να κάνουμε για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την δράση μας, δράση τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλία, κυρίως τώρα που είναι ε, Χριστούγεννα και πάρα πολλές τέτοιου είδους επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τον αθέμητο ε, συναγωνισμό και αθέμητο τρόπο δράσης ε, ενοχλούν τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ε, η δική μου τροπολογία να πω ότι είναι η 13, να την προσθέσετε στον κατάλογο τροπολογιών. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Η κυρία Σινάλοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μετά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν προηγουμένως και την ερώτηση που έγινε, δηλαδή είπαμε ότι σε μία προφορική τροπολογία θα μπορούσαμε να πούμε παραδείγματος χάρη διότι η αιτιολογική έκθεση της ε, Επιτροπής αυτό αναφέρει. Εάν μας αναφέρει κάποια παραδείγματα η Επιτροπή και τονίσει ότι πρόκειται μόνο για παραδείγματα, ίσως δεν θα χρειάζεται να κάνουμε πλήρη αναρρύθμιση. Εάν όμως αυτή η προσέγγιση δεν γίνει αποδεκτή από το ΕΛΚΑ, θα μπορούσαμε να βρούμε μια πιο γενική διατύπωση και να την υποβάλουμε στο ΕΛΚ σήμερα το απόγευμα. Θα πρέπει να δούμε ίσως μια πιο γενικότερη διατύπωση για να μην ε, αναφέρουμε μόνον, για να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα όπως σας είπα, για να μην έχουμε διεξοδικό κατάλογο. Σίγουρα Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και είμαστε ανοιχτοί σε μικροτροπολογίες, θα βελτιώσουν το όλο θέμα. Εάν όχι, θα δώσω τον ε, λόγο στον κύριο Γρίχο, ο οποίος εκ μέρους της Επιτροπής είναι από νομική πλευρά υπεύθυνο για να μα πει από τη δική του άποψη τι πιστεύουν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω και εσά και τον κύριο Χοσφόρ, ο οποίο επεξεργάστηκε αυτό το έγκαιρ Πάλι έχω ήδη πει πόσο τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε συνάδουν με τα δικά μας. Και αναφέρομαι στην ε, έκθεση του Μαρτίου 13 για την εφαρμογή της οδηγίας Πρέπει να πω ότι οι τροπολογίες και οι παρατηρήσεις που έγιναν ε, επίσης από την Επιτροπή σας και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων επίση συνάδουν με την ε, όλη άποψή μας και τα συμπεράσματά μας. Ήδη στο παρελθόν σχολίασα διεξοδικά τις παρούσες πρωτοβουλίες θα μπορούσα να τις συνοψίσω και να σας πω ποιες είναι οι δράσεις που αναλαμβάνουμε για να απαντήσω στα θέματα που θέσατε στη συζήτηση. Εδώ σε δύο τομείς επικεντρωνόμεθα. Πρώτα απ' όλα γενικότερα η εφαρμογή και η ανάγκη να ενισχυθεί η εφαρμογή αυτού του συστήματος και δεύτερον ιδιαιτέρως αναφέρομαι σε κάποιες ιδιαίτερες εμπορικές πρακτικές, κυρίως αυτές τις νέες πρακτικές ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου και νέες μορφές ε, ε, διαφήμισης και προσέγγισης των καταναλωτών. Το θέμα που μας απασχολεί πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι καταναλωτές. Τα παιδιά και η τρίτη ηλικία. Λοιπόν, η εφαρμογή. Ας επανέλθω στο πρώτο θέμα. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση της οδηγία και να έχουμε μία πιο στοχευμένη εφαρμογή. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να το κάνουν και τα κρατημέλη και να μπορέσουν στον συντονισμό αυτό που θα γίνει να ενισχύσουν και τις ε, ε, αρμοδιότητες της Επιτροπής. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία ελέγχθησαν σήμερα από τους συναδέλφους σας, στην έκθεση, στο πρώτο μέρος ασχολούμεθα με την, τον έλεγχο της εθνικής εφαρμογής, αν θέλετε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλοι κανόνες και η σωστή μεταφορά της οδηγίας στο κάθε εθνικό δίκαιο. Συνεχίζουμε. We have, we are a broad transposition Πώς γίνεται η μεταφορά μέσω ελέγχων, διαλόγου, ε, σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα, παραβιάσεις κτλ. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί λοιπόν. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε εδώ, συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών. Δηλαδή, αυτοί που εφαρμόζουν την οδηγία να μπορέσουν να την ενθαρμόσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όχι μόνο σε περίπτωση διαμεθοριακής συνεργασίας, αλλά για να προστατευτούν όλοι οι καταναλωτές. Τώρα, κάνουμε, όπως ξέρετε, με τις εθνικές αρχές διάφορα σεμινάρια για την εφαρμογή της οδηγίας και κυρίως ασχολούμεθα με συγκεκριμένες πρακτικές που αφορούν την αγορά σε διάφορα θέματα και η αναθεώρηση του κανονισμού για την προστασία των καταναλωτών επίσης είναι κάτι σωστό. Η ενίσχυση του όλου δικτύου για θέματα διασυνοριακά, τα οποία καταρχάς εγκρίθηκε η οδηγία, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Και όπως ξέρετε, η διαδικασία αναθεώρησης συνεχίζεται και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα έχει ολοκληρωθεί. Η ιδέα δεν είναι να βελτιωθεί σε θέματα διασυνοριακά συνεργασία, αλλά να προσπαθήσουμε, αν θέλετε, το δίκτυο να το επεκτείνουμε και πέραν. Δηλαδή, θέματα που αφορούν τους καταναλωτές, τους, ε, ε, την ευρύτερη ομάδα των καταναλωτών, πέραν από διάφορα τεχνικά θέματα διασυνοριακά και ελπίζουμε ότι επίσης και εδώ η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2014. Το τρίτο θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας, είναι ο οδηγός εφαρμογής της οδηγίας, διότι τα περισσότερα θέματα αφορούν από τελεσματικό τρόπο εφαρμογής της, που θα έγκυται στην σωστή ερμηνεία των κανόνων και ότι οι διεθνικές αρχές θα έχουν, θα εφαρμόζουν από κοινού όλους αυτούς τους κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το 2014 θα ενημερώσουμε αυτό το σχετικό έγγραφο τον οδηγό εφαρμογής και υπάρχουν επίσης κάποια θέματα που ανέφερε ο κύριος Ροσφόρ για την εκ των υστέρων ε, παρακολούθηση του όλου θέματος και από την Επιτροπή Νομικών θέματων τα το θέμα των κοινωνικών μέσων, τα θέματα των τιμών στον τομέα των ταξίδιων, διάφορες ε, διεκδικήσεις σε περίπτωση παράβασης και κυρίως θα ασχοληθούμε και με τους ευάλωτους καταναλωτές. Τώρα, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε σαφείς κανόνες όταν έχουμε να κάνουμε με επιθετικές ε, μορφές εμπορικών τέτοιων πρακτικών που αφορούν κυρίως τα παιδιά και τους μεγάλους ανθρώπους. Τα παιδιά, Φερρυπίν. Ένα θέμα που θα καλύψουμε είναι πώς θα μπορέσουμε να έχουμε νομική κάλυψη για τις διάφορες ε, online αγορές που γίνεται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με τα οποία παίζουν τα παιδιά γίνονται σχετικές ε, ε, μελέτες που θα διαρκέσουν 8 μήνες με στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες συστάσεις για τον τρόπο που θα λειτουργεί η αγορά. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι θα θέλαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή οι εθνικές αρχές και όλοι όσοι μας συνδράμουν για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό τον οδηγό εφαρμογής. Φερρυπίν, ε, σε θέματα σύγκρισης τιμών, σε θέματα περιβαλλοντικά. Έχει γίνει διάλογος που σχεδόν διήρκε σε ένα χρόνο με εκπροσώπους των εθνικών αρχών, ενώσεις καταναλωτών, εκπροσώπους της βιομηχανίας που προσπαθούν να εντοπίσουν τα κυριότερα προβλήματα και να κάνουν τις συστάσεις που αφορούν την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν. Και όλες οι παγιωμένες απόψεις στο τέλος θα συμπεριληφθούν σε αυτόν τον οδηγό εφαρμογής. Επίσης υπάρχει το αποθετήριο, η βάση δεδομένων αν θέλετε, που θα είναι στη διάθεση των πολιτών και θα αφορούν ό,τι αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές από την νομοθεσία, ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογής κτλ. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή την παρούσα βάση δεδομένων να την ε, συγχωνεύσουμε με μία καινούργια ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα, μία ενοποιημένη βάση δεδομένων για την προστασία των καταναλωτών. Πέμπτη παρατήρηση δίκτες εφαρμογής. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τους δίκτες επιδόσεων της κάθε χώρας όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιους δίκτες που θα μας επιτρέψουν να συγκρίνουμε τις επιδόσεις του κάθε εθνικού συστήματος και να αξιολογήσουμε, να εκτιμήσουμε σε ποιο μέτρο κάθε σύστημα ε, αποδίδει, αποφέρει αποτελέσματα. Ένα μέρος θα αφορά τις κυρώσεις. Και το θέμα αυτό βεβαίως έχει σχέση με το θέμα των ε, συλλογικών προσφορών οι οποίες, προσφυγών που, πρέπει να, ε, που θα γίνονται σε περίπτωση ε, απατών ή παραβίασης του όλου συστήματος. Ένα άλλο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το θέμα της σχέσης, όπως ελέγχθηκε και προηγούμενες ε, ε, συνεδριάσεις, της οδηγίας για τους καταναλωτές και του οδηγίας SCB. Ε, όσον αφορά το B2B, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση σύντομα που από τη μια θα ενισχύσει τους κύριους κανόνες που αφορούν ε, τις, ε, το αθέμητο εμπόριο και τι απάτε από τι οποίε μπορούν να αποφέρουν διάφορε επιχειρήσει, κυρίως οι μικρές, και θα βελτιώσουμε και του μηχανισμού συνεργασία, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνε αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη και τον διασυνοριακό χαρακτήρα κάποιων από αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Εκτός αν έχει κάποιος περαιτέρω Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα είπατε, μας δώσατε μια πλήρη εικόνα για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε ε, τις ε, διατάξεις. Έχουμε τις εκθέσεις ε, για πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν έχουμε τυπική συνέχεια, επίσημη συνέχεια εμείς και θα δείτε τι θα γίνει με το επόμενο κοινοβούλιο. Εμείς θα ψηφίσουμε αύριο και θα μπορέσει να, να αποτελέσει αυτό βάση για το επόμενο κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν εν ευθέτω χρόνο η ψηφοφορία διότι η Επιτροπή αυτή ήταν υπεύθυνη για την υιοθέτηση της αρχικής οδηγίας που ήταν ε, ριζοσπαστική, ε, επαναστακενοτόμος οδηγία που αφορούσε τα προβλήματα των καταναλωτών. Κύριε Ροσφόρ, θέλετε να λάβετε το λόγο πρωτού κλείσουμε το θέμα αυτό. Ναι, θα το κάνω πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Νομίζω ότι βλέπουμε πολύ καλά ότι συγκλίνουμε και όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση, οι τροπολογίες, οι συμβιβασμοί και αυτό ικανοποιεί όλους. Η τροπολογία ε, σχετικά με την πολιτική συμφωνία δεν έχουμε πλήρη ενότητα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Ευχαριστώ την Κομισιό που μας εξέθεσε λεπτομερώς το πρόγραμμα εργασίας για το θέμα αυτό. Η σημασία που αποδίδεται στους ευάλωτους καταναλωτές είναι κάτι που τονίστηκε παρόλο που η Κομισιόν πήγε πολύ μακριά στον τομέα αυτόν, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάθε φορά που προστατεύουμε έναν ευάλωτο καταναλωτή, προστατεύουμε το σύνολο των καταναλωτών, διότι ο κάθε καταναλωτής δυνητικά θα μπορούσε να γίνει μια μέρα ευάλωτος, τροτός καταναλωτής. Το μόνο στοιχείο συζήτησης που αναφέρθηκε από τους συναδέλφους και παραμένει επιτάπητος είναι ο, ο τρόπος σύνταξης της τροπολογίας 7 για την αιτιολογική σκέψη G Υπάρχουν ε, διάφορες εκτιμήσεις ανάμεσα στο ΕΛΚ και στους σοσιαλιστές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εξήγηση. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι ε, ε, είναι ένα ετσέτερα που είναι στο κείμενο. Ε, της ε, Επιτροπής. Είναι ένα σημείο ε, πάρα πολύ ευαίσθητο και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τα όσα συμβαίνουν σχετικά με τις πωλήσει κατοίκων και τις πωλήσει που γίνονται εκτός των εμπορικών ιδρυμάτων. Και ξέρουμε παντού αθέμητες εμπορικές πρακτικές που θα πρέπει να ανοιχνεύσουμε, να καταδιώξουμε και να παρεμποδίσουμε. Το πρόβλημα αναφέρεται σε αυτά που πρέπει να κάνουμε και μήπως δεν θα πρέπει να στιγματίσουμε έναν τομέα ή άλλους τομείς εάν δεν φαίνεται προφανές τους συναδέλφους σχετικά με τον, την τροπολογία συμβιβασμού με τροπολογία προφορική, δεν ξέρω αν είναι συμβιβασμού, ίσως μια μέρα γίνει ως εισηγητής. Αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ σας, θα πρότεινα να επανέλθουμε στην αρχική διατύπωση της τροπολογίας έτσι όπως είχε ε, προταθεί από εσά, κυρία Σεβέλοβα, που είναι μια τροπολογία όπου δεν υπάρχει αναφορά σε έναν κατάλογο τομέων, είτε έναν ενιαίο κατάλογο τομέων, είτε το γεγονός να έχουμε αναφορές, έχουμε μερικές ώρες για να δούμε αν μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε για τον τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που θα ικανοποιούσε τους πάντες. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε ακόμα μερικές ώρες για να μιλήσουμε γι' αυτό. Πολύ καλά. Περιμένουμε τι θα ψηφίσουμε αύριο αλλά βλέπουμε ότι η υποστήριξη της Επιτροπής είναι σαφής. Ίσως θα επιφέρουμε μερικές λεπτομερείς αλλαγές. Νομίζω ότι με αυτούς τους συμβιβασμούς μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά στην πολιτική στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περνούμε σε ε, μια άλλη ε, εισήγηση για την οποία θα ψηφίσουμε αύριο ή τον Ιανουάριο. Όχι, όχι, δεν είναι αύριο. Ε, πρόκειται για την πρόταση του συστήματος e-call σε οχήματα. Θα δώσω τον, λόγο στην κυρία Σενάλοβα. Ο κύριος Σβάπ θα μιλήσει εξ ονόματος του κύριου Βαντερκάμπ, ο κύριος Ροσφόρ εξ ονόματος του κύριου Μάντες. Η κυρία Ρούλε είναι εδώ και εγώ είμαι εδώ. Έχουμε λοιπόν τους, όλους τους ε, σκιώδες. Δίνω τον λόγο ε, στην κυρία Σενάλοβα για να σχολιάσει ε, τα, τις τροπολογίες και οι σκιώδεις και τα άλλα μέλη μπορούν επίσης να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Πετσινέλη είναι εδώ. Α, είναι εδώ, είναι εδώ. Είστε ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτος. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Κάρλο Πετινέλη θα δώσω το λόγο. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών εκπροσωπείται. Χαιρόμαστε πάντοτε όταν έχουμε εδώ τον κύριο Πετινέλη. Η κυρία Σενάλοβα, θέλετε να λάβετε το λόγο, να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση με, την, με, τις μεταφορές και ποια είναι η άποψη σας για τις τροπολογίες σχετικά με τους σκιώδεις εισηγητές νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ θετικές εδώ και 15 ημέρες και με την ευκαιρία αυτή διευκρινίσαμε τη θέση μας σχετικά με 123 τροπολογίες που λάβαμε. Συζητήσαμε επίσης με την Επιτροπή και νομίζω ότι δεν θα ήταν κακό να ομαδοποιήσουμε τις τροπολογίες σε ορισμένες κατηγορίες και να πούμε σαφώς ποια είναι τα περιεχόμενα αυτών των τροπολογιών και ποια είναι η, γνώμη μου εκ προημίου. Η πρώτη ομάδα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η ομάδα των προτάσεων που θα ήθελε να απορρίψουμε την πρόταση και που τονίζει την ε, προαιρετική ανάπτυξη, κυρία Ντε και άλλοι συνάδελφοι. Θα ήθελαν η ανάπτυξη της υπηρεσίας αυτής να είναι προαιρετική και απορρίπτουν το σύνολο της πρότασης. Εγώ ως εισηγήτρια πιστεύω ότι αυτό είναι αντιφατικό σε σχέση με το στόχο της πρότασής μου. Δεν πρόκειται λοιπόν να υποστηρίξω τις τροπολογίες αυτές και πολλές φορές ανέφερα ότι ο στόχος της εισήγησης αυτής είναι ε, να επανέλθουμε στην έκθεση πρωτοβουλίας που ήδη υιοθετήσαμε ως Κοινοβούλιο και όπου τονίσαμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτού του συστήματος ηλεκτρονικών κλήσεων. Η δεύτερη ομάδα τροπολογιών αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής και εδώ στην πρώτη φάση θα έλεγα ότι είμαι υπέρ της ανάπτυξης συστημάτων στα οχήματα, στα αυτοκίνητα, όπου υπάρχουν ήδη συστήματα κατάλληλα ενεργοποίησης. Κι όμως ορισμένοι συνάδελφοι είναι της γνώμης ότι θα ήταν καλό να καλέσουμε την Κομισιό να σκεφτεί επίσης για άλλες δυνατότητες, ούτως ώστε να παρουσιάσει μια πρόταση διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής αυτής της υπηρεσίας e-call για τις μοτοσικλέτες, βαρέα φορτηγά, ε, για τα πούλμαν, για τα λεωφορεία, αλλά επαναλαμβάνω άλλη μια φορά ότι σε μια πρώτη φάση θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στα συστήματα τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα. Θέση σε ισχύ. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζει μια άλλη ομάδα τροπολογιών. Όσον αφορά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ, οι προτάσεις ε, είναι διάφορες διστάμενες όσον αφορά τις δυνατότητες και τις προσεγγίσεις. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία τροπολογιών που θα πρέπει να εξετάσουμε. Οι συνάδελφοι Ροσφόρ και Χάμπρο προτείνουν 36 μήνες. Η κυρία Ρούλε προτείνει τον ε, Οκτώβριο 2017, δηλαδή 17 μήνες. Βαντεκάμπα προτείνει την προθεσμία των 17 μηνών, εγώ ως εισηγήτρια εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να ζητήσω από την ε, Κομισιόν μια ημερομηνία το 2015. Ε, με τον τρόπο αυτό απευθυνθήκαμε στην Κομισιόν και θελήσαμε η πρόταση αυτή να ισχύει για όλους τους νέους τύπους οχημάτων και επιμένω πάνω στην ημερομηνία αυτή του 2015, αλλά υπό ορισμένου όρους. Δηλαδή θα πρέπει να καλέσουμε το Συμβούλιο να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το σύστημα e-call, θα πρέπει η Κομισιόν να μπορέσει να προετοιμάσει όλες τις κατεξιοδότηση πράξεις που είναι μια προϋπόθεση απαραίτητη για την, ε, να προετοιμάσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία. Μια άλλη ομάδα τροπολογιών αναφέρεται στην ανοιχτή πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης και εδώ έχουμε αντιφατικές προσεγγίσεις, παραδείγματος χάρη ο κύριος Ροσφόρ, η κυρία Λεγκρίπ και άλλοι έχουν εξαλείψει την διάταξη για την ανοιχτή πλατφόρμα. Ο συνάδελφος Παντεκά Σαλβίνη, Χάμς και άλλοι αντίθετα τονίζουν ε, όλες τις διατάξεις σχετικά με την ανοιχτή πλατφόρμα. Ως εισηγήτρια είμαι της γνώμης ότι η ανάπτυξη όλων των άλλων εφαρμογών και υπηρεσιών επί του οχήματος δεν θα έπρεπε να καθυστερήσουν ε, την λειτουργία αυτού του συστήματος ή e-call που βασίζεται στο 112, αλλά ε, ε, βεβαίως η Κομισιόν θα πρέπει να εντείνει την εργασία της σχετικά με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίες που θα μπορούσαν να αποφέρουν ωφέλη για τους χρήστες, αλλά υπό τον όρο να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Μια άλλη ομάδα τροπολογιών αναφέρεται στην συνύπαρξη των ιδιωτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών που βασίζονται στον αριθμό κλήσης 112. Ο κύριος Βαντεκάπη, η κυρία Τούν και άλλοι συνάδελφοι, ο κύριος Χάρμπορ, μιλούν για ιδιωτικά συστήματα και τα βάζουν σε ίση μοίρα με τις δημόσιες υπηρεσίες. Πιστεύω ότι από την άποψη αυτή θα πρέπει να πούμε ότι η υπηρεσία η πανευρωπαϊκή που θα χρησιμοποιεί τον αριθμό 112 θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Βεβαίως μπορούν να υπάρχουν παράλληλα ιδιωτικές υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη συνέχεια για τους χρήστες. Θα πρέπει ε, να αποφύγουμε ιδιωτικές ε, υπηρεσίες να πάψουν να λειτουργούν όταν διασχίζουμε τα σύνορα. Θα πρέπει οι ιδιωτικές υπηρεσίες να έχουν κάποια συνέχεια. Έχουμε και το θέμα της προστασίας των προσωπικών ε, δεδομένων. Ο συνάδελφος Βάικελ Χέρτς προτείνει ο επιθεωρητής ο Ευρωπαίος και Καταναλωτών να τους συμβουλευόμαστε σχετικά με τις ε, κατάλληλες πράξεις. Υπήρξαν πολλές προτάσεις εκ μέρους της κυρίας Ρούλε για την ενίσχυση της σημασίας των ιδιωτικών, των προσωπικών δεδομένων. Συμφωνώ με την πρόταση αυτή. Θα πρέπει να πούμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ουσιαστική για τον τελικό χρήστη, αλλά θα πρέπει επίσης ε, να τονίσουμε ότι το σύστημα e-call δεν επιτρέπει ε, παρακολούθηση της κίνησης των ε, αυτοκινήτων. Αυτό πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Είναι ένα ε, σύστημα το οποίο κινητοποιείται όταν οι αισθητήρε των φουσκωτών μαξιλαριών αρχίζουν να λειτουργούν. Υπάρχουν ε, και άλλες τροπολογίες 73 εκεί όπου ζητούμε οι κατασκευαστές να αγγιηθούν η χρήση του e-call να επιτρέπει στους οδηγούς ε, να ακυρωσουν εκλίσεις εκκλήσεις e-call. Βεβαίως η βασική λειτουργικότητα του συστηματος η είναι να καλεί κανείς σε βοήθεια εκτάκτως το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει μια προφορική επικοινωνία όπου ο οδηγός μπορεί να δώσει εξηγήσει σε περίπτωση όπου το ατύχημα δεν είναι σοβαρό, που έχει τη δυνατότητα να μιλήσει, να εξηγήσει. Μετά υπάρχει η τροπολογία 80 του ιδίου συναδέλφου. Σε αυτήν την τροπολογία ε, ζητείτε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κλήσεις e-call χάρη στο σύστημα το νομαδικό των ε, κινητών τηλεφώνων και εδώ παραπέμπω στην έκθεση πρωτοβουλίας όπου τονίσαμε τα συστήματα επί των οχημάτων. Όσον αφορά τις ε, εγκαταστάσεις, τις νομαδικές, παρουσιάζουν πολλούς κινδύνους, διόπου μπορούμε να τον εξοπλισμό αυτό να τον αφαιρέσουμε, να ξεχάσουμε, ε, να τον ανοίξουμε, να τον θέσουμε σε λειτουργία. Πρέπει να επιμείνουμε πάνω στο σύστημα επί του οχήματος. Έχουμε και την τροπολογία 105 του ιδίου συναδέλφου που ζητάει οι χρήστες της υπηρεσίας αυτής να μπορούν να επενεργοποιήσουν ε, χειρονακτικά αυτή την υπηρεσία η call. Συζήτησα συχνά για το σύστημα αυτό, είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε ένα ε, δίθεν σύστημα ε, χάρη στους αερόσακους οι αισθητήρε, οι δέκτες μπορούν να θέσουν σε ενέργεια το σύστημα αυτό. Χαίρομαι που ορισμένε τροπολογίε αποσύρθηκαν, διότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων. Αυτές είναι οι παρατηρήσει μου για το ε, χειρονακτική απενεργοποίηση του συστήματος. Αυτό είναι ο κατάλογος των τροπολογιών που θα πρέπει να αναλύσουμε. Τώρα θα δουλέψουμε για την εκπόνηση συμβιβασμών και θα λάβουμε τις απόψει των άλλων επιτροπών. Χαίρομαι λοιπόν που θα μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με του σκιώδει Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που η κυρία Σενάλοβα σε πολλές περιπτώσεις υποστηρίζει αυτά που και εμείς ε, θεωρούσαμε προτεραιότητα ως ομάδα σε αυτήν την έκθεση. Ιδίως σε μια Ευρώπη που προστασία των δεδομένων αφορά για μας ένα μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων. Αυτό το τονίσαμε στις συνομιλίες των σχεδόν εισηγητών. Τώρα σήμερα μου ζητήθηκε να θίξω κάποια σημεία εξ ονόματος της σχεδόν συγκεντρίας μας. Ένα σημείο επιλήθηκε, διότι μπορεί η οδηγία να τεθεί σε ισχύ στην ημερομηνία που ανέφερε η κυρία Σενάλοβα. Είπε δυο λόγια για το θέμα αυτό, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε. Κατά δεύτερον, οι πτυχές προστασία των δεδομένων για μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το είπαμε και την, κατά την ακρόαση με τον κύριο Χάστινγκς. Το να υπάρχει από τη μία το σύστημα e-call και από την άλλη το e-safety είναι σημαντικό ώστε η προστασία των δεδομένων να διασφαλίζεται. Αυτό που θέλουμε και αυτό που μου ζητήθηκε να πω είναι το, ε, ο ενιαίος αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 να αρχίσει να ισχύει άμεσα σε όλα τα κάτι μέλη. Βέβαια το πρόβλημα είναι αν η Νορβηγία και η Ελβετία θα καλύπτονται. Ο κύριος Φάντενκαμπ είναι πεπισμένος ότι το σύστημα TPS μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και επιπλέον έχω και εγώ υποβάλει κάποιες τροπολογίες μαζί με την κυρία Δεγκρή για να υπάρχει μια καλή διάκριση μεταξύ των δύο συστημάτων. Μία πράσινη πλατφόρμα είναι ένα σημείο που δεν έχει ε, ακόμα συζητηθεί αρκετά. Υπάρχουν κάποιοι που συνηγορούν υπέρ ε, της πλατφόρμας, κάποιοι κατά, όμως για όσους ετοιμάζουν λογισμικά προτιμούν να υπάρχει ανοιχτή πλατφόρμα. Για να υπάρχει ένα κλειστό κύκλωμα στην ε, πλατφόρμα είναι λίγο δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια μέση οδός ώστε όσοι ήδη έχουν επενδύσει σε αυτά τα συστήματα να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Επιτρέποντας τους καταναλωτές να έχουν καλύτερη πρόσβαση. Υπάρχουν ακόμη κάποια σημεία που μου ζητήθηκε να δείξω. Το ποιε κατά τι πράξει θα περάσουν στα χέρια τη Επιτροπή και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Διότι στο κάτω-κάτω Δεν μπορεί όλα τα σημεία που είναι σημαντικά ιδίω για αυτή την ανοιχτή πλατφόρμα να εξουσιοδοτηθούν. Ίσως θα χρειαστεί μια επιπλέον οδηγία. Δεν μπορεί όλα να λυθούν εδώ. Ίσως όμως να χρειαστεί και κάποια διεύθυνση από την ε, Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν οι καλέ μα συνομιλίε και θα καταφέρουμε να βρούμε όλε τι απαραίτητε λύσει. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ που αναφέρατε όλα αυτά τα σημεία. Ο κύριος Φαρντανκάπ όντω είναι πολύ ενεργό στην προετοιμασία αυτού του κειμένου. Δεν είναι εδώ κανεί από του ε, φιλελευθέρου, η κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγητρία, η οποία τόσο καλά διοργάνωσε όλε τι συζητήσει των ε, σχεδόν εισηγητών, γιατί φτάσαμε στην ουσία του θέματο πολύ γρήγορα και καταφέραμε να επιλύσουμε τα προβληματικά σημεία. Σε ό,τι αφορά τη θέση σε ισχύ το 2017 ήταν αυτό που ζητήσαμε. Διότι το 2015 δεν είναι βέβαιη η ημερομηνία. Έχουμε αντικρουόμενες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για το κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό ή όχι. Θα είναι λοιπόν ε, διαφορετικές οι καταστάσεις από κάτω μέλος σε κάτω μέλος και καλό θα ήταν να παραμείνουμε εδώ ρεαλιστές. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Απλώς θέλω να σας το ρωτήσω για να δω αν ε, έχετε ε, λάβει υπόψη το τι διακυβεύεται. Για τις ε, τροπολογίες περί δεδομένων. Θα αποσύρουμε και την τροπολογία που σας δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά ο λόγος που τον είχαμε βάλει αρχικώς είναι γιατί και εμείς είχαμε κάποιες δυσκολίες. Όμως ετοιμάσαμε και ένα ενημερωτικό σημείωμα γι' αυτό διότι θέλαμε να είναι σαφή η διάκριση για την προστασία των δεδομένων μεταξύ του ε, ενιαίου αριθμού 112 και των επιπλέον ε, συστημάτων που θα προβλεφθούν. Τα ε, επιπλέον συστήματα θα τα παρέχουν ιδιωτικοί φορείς και αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Όμω, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα περισσότερα σημεία. Σα ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Νομίζω γρήγορα κάναμε. Ήταν σημαντικά τα στοιχεία που θίξατε. Και βεβαίω δεν μα διευκόλυνε στο να οδηγηθούμε σε γρήγορο πέρα τη εξέταση τη έκθεση και το τι έγινε στην Επιτροπή Λίμπερ. Μίλησε ο πρόεδρο τη Επιτροπή, νομίζω, εκεί για τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων. Εδώ όμω δεν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, μιλάμε για δεδομένα περί του οχήματο που διασφαλίζουν την ασφαλεία, ενεργοποίηση συστημάτων ασφαλεία σε οχήματα συζητούμε. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν κάποια, υπάρχει κάποια εμβολία για το αν το, θέμα θα το σύστημα θα πρέπει να είναι εθελοντικό ή όχι. Μίλησε κυρία Συνάλλοφα για τη δυσκολία που έχουμε με την ενεργοποίηση των αερόσακών σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν αισθητήρε ή όχι. Ε, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίε με τα παιδικά καθίσματα λόγου χάρη, με το ποιε θέσει επιβατών θα έχουν ε, αερόσακου και πώ θα ενεργοποιούνται ή όχι οι αερόσακοι. Ε, υπάρξ, υπήρξαν πολύ σοβαρά ατυχήματα. Κάποιοι έχουν χάσει τι αισθήσει του από μακρισμένε περιοχέ και βεβαίω αυτό εφόσον συμβεί θα πρέπει να ε, αποστέλνει ένα σύντομο σήμα, ένα πολύ γρήγορο σήμα για τη φύση του ατυχήματο και για το γεωγραφικό εντοπισμό του. Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλώς ποιος είναι ο κάτοχος του οχήματος, αλλά ποιος επιβαίνει στο όχημα. Άρα το σύστημα αυτό ε, για την ώρα δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα, αν όμω κανένα αρχίσει να προσθέτει δεδομένα, μπορεί και να λάβει πιο προσωπικό χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν με την κυρία Ρούλε να το δείτε κυρία Σενάλοβα για να βεβαιωθείτε ότι προχωρά το θέμα και συμφωνείτε και κάποιες από τις ε, υπηρεσίες που προσφέρονται από κάποιους απαρόχους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως υποκατάστατο. Έτσι, ώστε ως προς τα δεδομένα να καλύπτονται όλες οι εγγύσεις και να παραμένουν τα δεδομένα ανώνυμα πέραν των όσων αφορούν το όχημα. Όμω νομίζω ότι με την δουλειά που θα κάνετε θα μπορέσετε να καταλήξετε σε κάποια εικονοποιητική διατύπωση. Ω προ τα υπόλοιπα σημεία μπορώ να συμφωνήσω. Διότι νομίζω το πλέον σημαντικό είναι εδώ να έχουμε μια ρεαλιστική ημερομηνία ώστε όντω να πετύχουμε αυτό που επιδιώκουμε. Το πρόβλημα βεβαίω είναι ότι εδώ μιλάμε για περίπλοκα συστήματα. Το αναφέρει και ο κύριο Πέτερη. Ε, δεν μιλάμε για το ότι θα κάνει απλώ η αυτοκινητοβιομηχανία που καθορίζεται το οχήματο, αλλά η αποτελεσματικότητα του συστήματο ώστε να πετύχει τα αποτελέσματα που επιδιώκει ω προ την ασφάλεια και τη βελτίωση τη ασφάλεια, τη μείωση των ε, τραυματισμών και των ατυχημάτων, αυτό έχει να κάνει με το σύνολο του συστήματος, δηλαδή ακόμα και με τα συστήματα απόκριση ε, τα, το δημόσιο τομέα ή τη δυνατότητα του δικτύου να αντέξει το σύστημα, αλλά και το κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα προβλέψουν συστήματα επικοινωνίας που να συνδυαστούν απευθεία με τις ε, υπηρεσίε τους για τα επίγοντα. Είναι μια σειρά δηλαδή από διαφορετικούς φορείς που θα εμπλακούν στην όλη διαδικασία και διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών συστημάτων που πρέπει να γίνουν σωστά. Δεδομένου ότι όλα αυτά θα έχουν να κάνουν αποκεντρωμένες αρμοδιότητες για τοπικούς ή αποστάσεως ε, παρέχοντες υπηρεσίες, το σύστημα που οικοδομούμε είναι αρκετά περίπλοκο. Γι' αυτό και η δική μου τροπολογία. Νομίζω ότι 36 μήνε ήταν ένα λογικό διάστημα ώστε να μπορέσει να λειτουργεί επαρκώ ολόκληρο το σύστημα. Όμω, επειδή δεν μπορούμε απορριτήτω να δημιουργήσουμε προσδοκίε στου καταναλωτέ και μετά να του απογοητεύσουμε, θα πρέπει να προσέξουμε. Θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε περαιτέρω. Τώρα, κοιτάζοντα τι τροπολογίε, νομίζω ότι αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι σε γενικές γραμμές οι τροφολογίες μοιάζουν, δηλαδή είδα ότι οι δικές μου τροπολογίες μοιάζουν με κάποιες από αυτές των συναδέλφων. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποια σημεία σύγκλησης και απόκληση ταυτόχρονα, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι είναι το πιο λογικό να κάνουμε. Σίγουρα η κυρία Συνάλογα με την ε, πείρα που διαθέτει θα μα ε, βοηθήσει καθώ και όλοι οι υπόλοιποι σκέφτε εισηγητές, όπω έχει γίνει ως τώρα. Νομίζω λοιπόν ότι γρήγορα θα καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα με όλα αυτά. Τώρα, πριν καλέσω τον κύριο Πετινέλη να μας δώσει τη δική του άποψη. Ήθελα να δω αν κάποιος από τους συναδέλφους ήθελε το λόγο. Κάποιος άλλος. Ξέρω το παρακολουθείτε στενά το θέμα, γι' αυτό και σας άφησα χρόνο. Πρόεδρε, εάν θέλετε να σχολιάσω, συγχαίροντας την κυρία Σενάλοβα για την εξαιρετική της δουλειά, και για το πνεύμα συνεργασίας που πέδειξε. Διότι πράγματι καταφέρατε να, ε, κρατήσετε, να κρατήσετε τις σημαντικότερες, τις σοβαρότερες προτάσεις από όλους τους γύρους συνομιλιών που είχαμε. Επικεντρωθήκατε στο να βρείτε την ε, άριστη η πιο εύστοχη λύση και μάλιστα όσο δυνατόν συντομότερα. Γι' αυτό κοιτάζουμε προσεκτικά το τι συμβαίνει και στα επιμέρους κράτη-μέλη και θα πρέπει να δούμε αν εφαρμόζουν το σύστημα του ενίου αριθμού, του 112. Έχουμε σοβαρέ αμφιβολίες εδώ. Συζητήθηκε επανειλημμένος και το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί. Δεν λειτουργεί πάντοτε όμως ε, στην προσωρινή του φάση όπως θα έπρεπε. Παραμένουν λοιπόν προβλήματα και σίγουρα θα παραμένουν και στο μέλλον, είτε το 2015 είτε το 2017. Να τονίσω τα εξή δύο τώρα. Ότι βεβαίω επιδιώκουμε την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και θέλουμε να υπάρχει ελευθερία στην επιλογή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια όμως. Όλο και περισσότερα στοιχεία γίνονται ε, υποχρεωτικά. Ακόμη συζητούμε τους αεροσάκους, τις ζώνες ασφαλείας, τα κράνη που έχουν γίνει πλέον ε, υποχρεωτικά για τους ε, οδηγούς μηχανοκινητών δικύκλων το ίδιο και για αυτό το σύστημα. Το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να απενεργοποιείται. Εάν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίηση ή εγκατάστασή του σε κινητέ συσκευέ, δεν θα λειτουργεί όπω πρέπει. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπινε ζωέ. Κάποιε συσκευέ διασφαλίζουν την προστασία των ταξιδιωτών και έχουν συζητηθεί πολύ στο παρελθόν. Αλλά εδώ μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπινες ζωές ετησίως και το σύστημα αυτό θα πρέπει να λειτουργεί υποχρεωτικά, όχι να είναι αντικείμενο επιλογής. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανείς? Ωραία. Κύριε Κάρλο Πετινέλη, παρακαλώ να σχολιάσετε και μετά θα δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Σενάλογα για να ανακεφαλαιώσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή ΙΜΚΟ και την εισηγήτρια, την κυρία Σανάλοβα, διότι θεωρούμε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά για το φάκελο αυτό, διότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ζήτημα. Μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βασικά κεφάλαια, δηλαδή ομάδες τροπολογιών, όπως υποβλήθηκαν από την εισηγήτρια. Πρώτο, δυνατότητα εθελοντικής χρήσης του συστήματος e-call. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς δεν συμφωνεί με την πρόταση αυτή, διότι θεωρούμε ότι το να γίνει το σύστημα προαιρετικό θα αποδυναμώσει τα ωφέλη ασφαλείας του συστήματος. Για κάθε συσκευή ασφαλείας στο όχημα θα πρέπει να είναι ενεργή Εκτό αν υπάρχουν ειδικέ ανάγκε των επιβατών. Δεν θα πρέπει να μπορεί να απενεργοποιείται όμω η συσκευή γιατί μιλάμε για ασφάλεια και θα μειώσουμε πολύ σημαντικά το επίπεδο ασφαλεία. Αυτό που θέλουμε, ο στόχο τη πρόταση αυτή είναι να προσφέρει σε όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση τι ίδιε ταχείες και άμεσε αποκρίσει σε κατεπήγουσες ανάγκες σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματο. Δεν θέλουμε λοιπόν να μπορεί να απενεργοποιείται το σύστημα. Δεύτερη ομάδα τροπολογιών για το πεδίο της πρότασης. Εδώ υπήρξαν τροπολογίες για την διεύρυνση της ε, χρονικού χαρακτήρα του συστήματος αυτό. Πέραν των κατηγοριών που καλύπτονται αυτή τη στιγμή από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε ακόμη και άλλα να καλύψουμε. Αλλά το 90% των νέων οχημάτων λογικά καλύπτεται. Οπότε, θεωρούμε ότι η μελέτη αντικτύπου και η ανάλυση των πολλαπλών αποτελεσμάτων που ούτω ή άλλω χρειάζεται για οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση είναι κάτι το ε, που υπάρχει και ήδη διαθέτουμε για αυτά τα οχήματα. Τα δεδομένα λοιπόν που έχουν χρησιμοποιηθεί από την πλευρά της Επιτροπής με παράδειγμα τα μηχανοκίνητα δίκυκλα θα πρέπει να έχουν το δικό του σύστημα για την ε, ειδοποίηση σε περίπτωση ατυχήματο. Καλύπτουμε λοιπόν όσα περισσότερα γίνεται, αλλά κυρίως τις περισσότερες ομάδες οχημάτων. Η δεύτερη ομάδα τροπολογιών αφορούν τη θέση σε ισχύ και την ημερομηνία θέση σε ισχύ. Βεβαίω η θέση σε ισχύ θα εξαρτηθεί από την έγκριση της πρότασης και δευτική, γιατί η νομοθεσία θα εφαρμόζεται μόνο σε νέους τύπους οχημάτων. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε τις, ε, να παραμείνουμε πιστοί στην τωρινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι από αυτήν την ημερομηνία και μετά θα εφαρμόζεται η οδηγία στους νέους τύπους οχημάτων και όχι στους παλιούς για να καλύπτονται τα πάντα από την οδηγία αυτή καλό θα είναι να παραμείνουμε στην αρχική πρόταση της ε, Επιτροπής. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι πιέζει κάπως ο χρόνος για την προετοιμασία του συστήματος. Μια άλλη ομάδα τροπολογιών αφορά την ανοιχτή πλατφόρμα πρόσβασης. Η ε, πλατφόρμα αυτή διαφέρει κάπως από το σύστημα Equal. Δηλαδή η πρόταση όπως την έχετε επικεντρώνεται στο συστημα η e-call και τον ενίο αριθμό 112 ε, για τα κατεπήγοντα. Η άλλη εναλλακτική, η πλατφόρμα ανοιχτή πρόσβαση. Ναι, ναι, βεβαίω είμαστε πρόθυμοι να το συζητήσουμε. Όμω θα χρειαστεί διαφορετική μελέτη αντικτύπου και διαφορετική εξέταση του όλου θέματο. Θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα. Οπότε θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόταση ω έχει και να επικεντρωθούμε μόνο στον ε, αριθμό ε, ανάγκη. Αυτό και για τον υπηρεσία TPS. Και αυτό διαφέρει από τον ενίο αριθμό. Θα χρειαστούν πιο εξελιγμένες συσκευές από ό,τι για το σύστημα e-call όπως το προτείνουμε και εδώ πιστεύουμε ότι χρειάζεται διαφορετική εξέταση και διαφορετική πρόταση ενδεχομένως. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, το θέμα της προστασίας των δεδομένων είναι κάτι διαφορετικό, διότι το 112 είναι ανώνυμο σύστημα. Δεν μεταδίδονται πληροφορίες εάν δεν ενεργοποιηθεί το σύστημα. Είναι διαφορετικό να έχει κανείς ένα σύστημα, ένα κινητό, μια κινητή συσκευή στην τσέπη του και να την απενεργοποιεί στο όχημα. Με το σύστημα προτείνουμε είναι κανείς συνέχεια ε, ε, συνδεδεμένος. Είναι διαφορετικά λοιπόν τα πράγματα από την πλευρά της ε, προσωπικής ασφάλειας. Έχουμε την οδηγία 9136 που καλύπτει το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Οπότε αν αρχίσει να ισχύει η οδηγία αυτή και χρειαστεί να αναθεωρηθεί η οδηγία περί προσωπικών δεδομένων, προφανώς θα αναθεωρηθεί αναλόγως και η οδηγία ECOL για να λάβει υπόψη τις νέες προδιαγραφέ για την προστασία των δεδομένων. Η τελευταία ομάδα τροπολογιών αφορούν τα κινητά τηλέφωνα. Νομίζουμε ότι η λύση αυτή δεν αρμόζει για τις ανάγκες ασφάλεια που θέλουμε να καλύψουμε και για όλους τους λόγους που ανέφερε και η Συγγήτρια. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Οι συσκευές αυτές δεν προσφέρουν καμία εγγύηση ότι θα λειτουργήσουν εάν υπάρξει μια επίγουσα κλίση. Αυτό συμβαίνει γιατί υπήρξε μια σοβαρή σύγκρουση, ένα τύχημα που ενεργοποίησε τον Ρώσακο. Εάν έχει κανείς μια κλασική συσκευή κινητού, όπως ένα iPhone κάπου στο αμάξι του, στο αυτοκίνητό του, δεν σημαίνει ότι αν υπάρξει σύγκρουση θα λειτουργεί αυτό. Μπορεί να σπάσει, μπορεί να καταστραφεί. Νομίζω ότι λίγο πολύ κάλυψα τις περισσότερες τροπολογίες, ανακατηγορία. Σταματώ λοιπόν εδώ με τα σχόλιά μου και είμαι στη διάθεσή σας από όσων υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την συνολική παρουσίαση και κάλυψη των θεμάτων. Νομίζω όντω κάλυψατε όσα σχολίασαν και οι συνάδελφοι. Θέλει κάποιο να δευτερολογήσει, ή να λόγω το λόγο στην κυρία Σενάλογα για να σχολιάσει τα όσα ακούστηκαν και να μας πει και ποια είναι τα επόμενα βήματα βάσει του χρονοδιαγράμματος. Ίσως να μας επιβεβαιώσετε και πώς προχωρά ή να μας ενημερώσετε για το πώς προχωράει η Επιτροπή Μεταφορών εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδελφούς για τα θετικά τους σχόλια και για τις συνεισφορές τους. Νομίζω ότι λίγο πολύ συγκλίνουμε στις απόψεις μας. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έδωσε τη γνώμη της ανακατηγορία τροπολογιών ως εισηγήτρια οφείλω να διαπιστώσω ότι συμφωνώ με το σύνολο των σχολείων που ακούσαμε. Συνειδητοποιώ ότι το θέμα της ημερομηνίας θέση σε ισχύ είναι ένα θέμα που θα πρέπει να λυθεί. Να λυθεί με τρόπο ε, ρεαλιστικό. Από τη μια, εδώ είχαμε το θέμα της ταχείας, ε, είχαμε μάλλον την επιλογή της ταχείας προσέγγισης και από την άλλη υπάρχει και η ανάγκη να ετοιμάσουμε ένα σύστημα τέτοιο που να είναι τελείως αξιόπιστο και να λειτουργεί. Δηλαδή δεν μπορεί το Κοινοβούλιο μόνο του να αποφασίσει για την ημερομηνία. Υπάρχουν και οι υπόλοιποι συνομιλητές μας, ε, κατεξοχήν το Συμβούλιο, Και εκεί πραγματικά βασίζω τι ελπίδες μου στην ελληνική προεδρία που είπε ότι το σύστημα θα είναι μια από τις προτεραιότητές τη στον τομέα των ε, μεταφορών. Εάν λοιπόν θελήσουμε να επιταχύνουμε την εισαγωγή του συστήματος αυτού, θα πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι μας χρειάζεται να έχει θετική στάση και το Συμβούλιο. Τώρα, ε, η Επιτροπή μίλησε για τον Οκτώβριο του 2015 και είπε ότι η ημερομηνία αυτή φαίνεται ρεαλιστική. Εγώ θέλω να παραμείνει η ημερομηνία αυτή στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι το αν θα προκριθεί αυτή η ημερομηνία ή όχι εξαρτάται και από το πώς θα λυθεί το θέμα των κατακρισουσιοδότηση πράξεων και ούτω καθεξής. Σε αυτή λοιπόν ακριβώς τη χρονική στιγμή δεν έχω κάτι καλύτερο να προτείνω, πέραν των όσων είχα προτείνει στην αρχική μου τροπολογία, σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα, την ανοιχτή πλατφόρμα. Συμφωνώ με εκείνον που είπε ότι η ανοιχτή πλατφόρμα θα πρέπει να είναι αντικείμενο ξεχωριστού νομοθετήματος. Άλλωστε, είπα, αυτό δεν είναι η και του τροπολογίε μου, η και βεβαίω συμφωνώ. Συμφωνώ ότι η προστασία των δεδομένων πρέπει να διασφαλίζεται πλήρω. Και μάλιστα έτσι, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσει, ώστε να μην ε, μπορεί να υπάρξει κερδοσκοπία ως προς τα οχήματα. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα και το πώς θα προχωρήσουμε. Σήμερα συζητιέται το θέμα στην Τραν. Αύριο η Επιτροπή μας θα ψηφίσει για την ε, έκθεση αυτή. Ε, στις 9 Ιανουαρίου η Επιτροπή Ήτρε. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι θα κάνει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όμως για τη δική μας Επιτροπή προκύπτει ότι θα δούμε τις τροπολογίες στις 22 Ιανουαρίου, 22 Ιανουαρίου και 23 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε. Του χρόνου εννοείται. Είμαι πλήρως πεπισμένη ότι την έκθεση αυτή την έχουμε συντάξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι θα έχουμε και ευρεία στήριξη από τους συναδέλφους. Η συνεργασία με, τις, με τους κοιόδης εισηγητές και εισηγητές ήταν εξαιρετική και νομίζω ότι θα πετύχουμε. Θα πετύχουμε να περατώσουμε την έκθεση αυτή εγκαίρως και ότι θα προλάβουμε να την εγκρίνουμε και εντός της δικής μας θητείας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Νομίζω ότι όντω πρέπει να στοχεύσουμε στις 23 Ιανουαρίου. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών μας είπε ότι θα ψηφίσουν στις 9 Ιανουαρίου. Εάν δεν ψηφίσουν εγκαίρως, αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένουμε και τη δική του ψηφοφορία, αλλά δεν βλέπω να υπάρξει λόγο να γίνει αυτό, γιατί ήδη έχουμε συνομιλήσει εντατικά για το θέμα τη εκτιμένης πρόταση. Θα το ξανασυζητήσουμε με τον πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα για να το καθυστερήσουν. Θα φροντίσουμε πάντω να δούμε πώ θα προχωρήσει και η δική του δουλειά για να συντονιστούμε. Ξέρω ότι και με τον ε, εισηγητή τη Επιτροπή Τραν έχετε ε, συζητήσει συχνά, γιατί χρειαζόμαστε και τη δική του στηρίξη για να λειτουργήσει το όλο δίκτυο. Πρέπει η όλη διαδικασία να ε, είναι συνολική και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Σενάλοβα για την τεράστια δουλειά που έχει κάνει εδώ και ε, σε συνεργασία με τα μέλη τη δική μα Επιτροπή και τη Επιτροπή Μεταφορών. Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στην επόμενη πρόταση, σε αυτή την τόσο φορτωμένη μερίσια διάταξη του σημερινού απογεύματο. Ε, τροπολογίε της για την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Νομισματικών Υποθέσεων και τους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Εισηγητής της Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων είναι ο κύριος Βαμπ. Τον έχουμε εδώ σήμερα το απόγευμα μαζί μας. Είμαι βεβαίως ότι θα σχολιάσει και από τη δική του σκοπιά την έκθεση αυτή και ο κύριος Σμιτ είναι εισηγητή από τη δική μα Επιτροπή. Έχουμε τέσσερι συμβαστικέ τροπολογίε που έχουν μοιραστεί στα μέλη. Φαντάζομαι ότι θα τι ε, θίξει ο κ. Σμιτ. Και μετά έχουμε τον κ. Σφάπ, την κυρία Ράπτη, την κυρία Ρούλε. Ε, το συνάδελφο Φόξ επίσης ε, με τον οποίο συνεργαζόμαστε για το θέμα αυτό ε, μου έχει αφήσει τις δικές του απόψεις για τις συμβαστικές τροπολογίες θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως δίνω το λόγο στον κύριο Σκουμί ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Αρχίζοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που προαναφέρετε δεν θα τους το επαναλάβω λοιπόν διότι με βοήθησαν για να καταλήξουμε σε συμβιβαστική πρόταση. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα. Και πολλές φορές ξέρω ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις και συζητήσαμε πολλά θέματα με του συναδέλφου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σμπάμπ. Ξέρω ότι είναι δικηγόρο. Εγώ είμαι απλό πολιτικό. Και πολλέ φορέ τέλο πάντων, στη συγκεκριμένη περίπτωση καταλήξαμε σε πολύ καλή συμβιβαστική λύση. Το έχω αναφέρει πολλές φορές και επαναλαμβάνω ότι πιστεύω ότι όντως είναι σημαντικό αυτό το θέμα και ίσως στην Επιτροπή μας θα μπορούσαμε να έχουμε και μία άλλη άποψη και να την εκφράσουμε όταν και στην ΕΚΟΝ θα εξεταστεί η εκθεσή σας. Είμαστε στην Επιτροπή μας υποχρεωμένοι να εστιαστούμε στα θέματα που αφορούν τους καταναλωτές Και Νικότερα πιστεύω εγώ ότι αν η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ολοκληρώσουν αυτή την περίφημη ενιαία εσωτερική αγορά, θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω στο συγκεκριμένο θέμα αυτό, διότι έχουμε σοβαρά προβλήματα και μπορώ να το καταλάβω το, και το καταλάβω. Είχαμε και στο παρελθόν σημαντικά προβλήματα, αλλά τώρα πλέον δεν έχουμε πολύ χρόνο στη θέση μας και δεν μπορούμε να χρονοτριβούμε αν δεν κάνουμε κάτι σωστό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί με τους κατάλληλους κανονισμούς και την κατάλληλη νομοθεσία η ενιαία εσωτερική αγορά. Κάναμε κάποιες συμβαστικές λύσεις. Πρώτα απ' όλα για τις συλλογικές ε, πρόσφυγες. Ίσως αυτό ήταν το πιο επίμαχο θέμα. Και πιστεύω ότι το κείμενο έτσι όπως τροποποιήθηκε θα βοηθήσει να γίνουν σωστά οι αποζημιώσεις για τους καταναλωτές με δίκαιο τρόπο και νομίζω ότι καταλήξαμε σε λύση την οποία πεδέχθησαν οι πάντες. Στην δεύτερη συμβαστική λύση επιτρέπουμε και σε όλα τους ε, κρίκους, αν θέλετε, της όλης αλυσίδας, να έχουν κάποια ε, αποζημίωση. Έχουμε προβλέψει την ε, ε, επιπλέον επιβάρυνση. Δεν θέλουμε να υπάρχουν διπλές αποζημιώσεις. Τρίτη συμβιβαστική λύση. Συζητήσαμε ε, και δεν ξέρω μπορούμε να συμφωνήσουμε, βαθέων κάποια πράγματα. Για μένα το 95% των καρτέλ δημιουργούν πρόβλημα. Βλάπτουν. Δεν ξέρω αν και εσείς το πιστεύετε πρόεδρε και δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε ότι γενικότερα τα καρτέλ ε, δημιουργούν πρόβλημα. Για μένα αυτές οι συμπράξεις, τα καρτέλ, ε, είναι ένας άσχημος όρος. Άσχημη λέξη. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι αυτή η συμβαστική λύση την οποία καταλήξαμε είναι λογική. Ώστε να μπορεί κανείς με λογικό τρόπο να εγείρει μια αξίωση αποζημίωσης και να αποζημιωθεί στο τέλος. Και ελπίζω ότι αύριο στην ψηφοφορία θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για να ε, πάει η γνωμοδοτή στην ΕΚΟΝ. Και βέβαια ο κύριος Σφάμπ να αλλάξει καπέλο να φορέσει ίσως ε, κάποιο άλλο όταν θα πρέπει να ληφθεί απόφαση στην ΕΚΟΝ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ πιστεύω ότι είμαστε εδώ για να προσπιστούμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και ευθύς εξ αρχής, ε, από τότε που είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαι της άποψης ότι όντως χρειαζόμαστε κάποια συλλογική δράση με λογικό τρόπο, με σωστό τρόπο, όχι άλλα αμερικάνικα. Και ελπίζω ότι αυτό θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε αύριο. Αυτό προσπάθησα να κάνω με τις συμβαστικές ε, τροπολογίες οποίες καταλήξαμε. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία όλων και πάντα είναι ενθαρρυντικό να ξέρει κανείς ε, ότι παρά το γεγονός ότι διαφωνεί με τη συζήτηση μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία. Και το αντίθετο βεβαίως μπορεί να συμβεί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος ο Αντρές Σφάμπ τώρα. Με τα δύο του καπέλα. Εισηγητής και σκιώδης εισηγητής σύγχρονος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως το είπατε κι εσείς προηγουμένως, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σμιτ και τους άλλους συναδέλφους, διότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και στέλνουμε ένα επικοδομητικό και σαφές μήνυμα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ που νομίζω ότι μας φέρνει πιο κοντά στις θέσεις όλων Και βεβαίως δεν θα πρέπει να θέσουμε σε αμφισβήτηση αυτό τον επικοδομητικό διάλογο με διάφορες επικρίσεις. Ο κύριος Σμιτ, συγγνώμη, η Επιτροπή μας γνωμοδοτεί στην ΕΚΟΝ ώστε να υπάρχει οι ίδιοι κανόνες και να εφαρμόζει το ίδιο δίκαιο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσπαθήσουμε να έχουμε μια δίκαιη μεταχείριση για όλους όσους υφίστανται ζημίες από κάποιο καρτέλ, από κάποια δημοσία. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια θέματα που μπορούν να βελτιωθούν ίσως από την νομική οπτική γωνία. Αλλά ούτως ή άλλως οι κανόνες που ανέφερε ο κύριος Σμιτ δεν έχουν μόνο ε, πολιτική χρειά. Πρέπει να δούμε από νομικής πλευράς πώς εδράζονται. Δηλαδή πρέπει να δούμε τη νομική βάση, πρέπει να δούμε ποια είναι η διαδικασία, τα μέτρα και το βάρος της απόδειξης βεβαίως. Η ζημία που υπέστη κάποιος όταν αξιώνει κάποιος αποζημίωση. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε προσεκτικά. Διότι εάν υπάρχει σύγχυση πρέπει να δοθούν αποδείξεις σαφείς. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Εν πάση περιπτώσει για την συμβιβαστική πρόταση 1... Δεν θέλουμε ποινή, αν θέλετε. Απλώς θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί κανείς, εάν εγείρει μία τέτοια αγωγή αποζημίωσης, να μπορέσει να αποζημιωθεί. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα κάποιες από τις τροπολογίες μου να τις ε, κρατήσω παρά το πολιτικό μήνυμα. 72, 73, 75 και θα δω και κάποιες άλλες. Κάποιες τις έχω αποσύρει έχοντας συζητήσει με συγητή, διότι πιστεύω ότι το, πολιτικό, το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε πρέπει να είναι πολιτικής χρειάς. Ε, και αύριο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ψηφοφορία. Τώρα με το άλλο μου καπέλο. Ελπίζω ότι θα μπορέσει το κείμενο αυτό να περάσει κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας ακόμη, πράγμα δύσκολο. Άρα θα πρέπει να επιδείξουμε μεγάλο συνενετικό πνεύμα όλοι μας. Και αύριο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα δούμε τι θα κάνουμε. Η γνωμοδότηση Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων θα είναι έτοιμη στις 21 Ιανουαρίου. Στην ΕΚΟΝ θα γίνει ψηφοφορία στις 27. Και αν καθυστερήσουμε, δεν θα μπορέσουμε την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου να κάνουμε το διάλογο μεταξύ των τριών μερών, άρα δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση στη διάρκεια της μας Κάνω θα ήθελα λοιπόν όλοι με πνεύμα λογικής να προχωρήσουμε σε αυτή την ε, συμβιβαστική λύση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας. Εγώ θα το κάνω αυτό με όλη την καλή θέληση και ελπίζω ότι και όλοι οι συνάδελφοι το ίδιο θα κάνουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ράπτη, το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτον να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σμίτ Προσυπογράφω απολύτως την εισήγηση που έκανε. Ήταν καθοριστική και καταλητική η δουλειά που έκανε και η συνεργασία που είχε μαζί μας για να φτιαχτεί η, αυτή η γνωμοδότηση. Ε, τώρα, ο κύριος Βάμπ έβαλε και με τα δύο καπέλα, εν πάση περιπτώσει, Ξέρετε, όταν έχει δύο καπέλα είναι πιο εύκολο. Εμεί έχουμε ένα καπέλο. Με αυτό πρέπει να βολευτούμε. Εν πάση περιπτώσει με τα δύο καπέλα ε, έβαλε, μας έβαλε εδώ μπροστά μα και το μαστίγιο και το καρότο. Και λέω και το μαστίγιο και το καρότο διότι από τη μια μεριά μας είπε ότι είναι πρόθυμος να ε, κάνει το καλύτερο δυνατό να αποσύρει και κάποιες τροπολογίες κλπ. Αλλά από την άλλη μεριά μα είπε ότι κοιτάξτε να δείτε αν θέλετε να ψηφιστεί ε, την τρέχουσα νομοθετική περίοδο η γνωμοδότηση αυτή, η έκθεση αυτή ε, πρέπει να συντομεύουμε, πρέπει να συμβιβαστούμε και αυτή είναι η κατάσταση. Ε, το κατανοώ, αλλά έχω στο μυαλό μου πάντα αυτό που υπογράμμισε ο κύριος Σμιτ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δουλεύουμε και να έχουμε στο μυαλό μας εδώ στην Επιτροπή μας την προστασία των καταναλωτών. Και επαναλαμβάνω και εγώ αυτό που είπε ο κύριος Σμιτ. Ε, τα καρτέλ κατά 95% ίσως και περισσότερο δεν κάνουν καλό στην υγεία των καταναλωτών. Κάνουν καλό στην υγεία των επιχειρήσεων. Εμείς πρέπει, έχουμε ε, ε, καθήκον μέγιστο να φροντίσουμε τους καταναλωτές, οι οποίοι ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα σε εποχές ε, κρίσης όπως αυτές που περνάει η Ευρώπη. Ε, τώρα για να μην είμαι άδικη, θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει πολλά θετικά στοιχεία. Ποιο είναι το μεγάλο έλλειμμα που έχει για τη δική μας άποψη, για τη δική μας πολιτική, το δικό μας πολιτικό γκρουπ. Ε, δεν προβλέπει το υποχρεωτικό collective redress. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, προχωράμε. Ο κύριος Σμίτ έκανε τέσσερις συμβιβαστικές τροπολογίες. Τις δεχόμαστε και τις τέσσερις. Είναι εξαιρετική δουλειά. Ωστόσο, υπάρχουν δύο σημεία που για μας έχουν χρώμα κόκκινο. Το λέω περιγραφικά, δεν το λέω κόκκινη γραμμή, γιατί οι δύο λέξεις κόκκινη γραμμή είναι πιο έντονες, πιο εμφατικές. Δείχνουν ίσως μια διαλαξία. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε πολύ πολύ σταθεροί στις γραμμές μας πάντα υπέρ των καταναλωτών. Έτσι λοιπόν ε, η μία περιοχή, να το πω έτσι, άντε να το πω γραμμή κόκκινη, είναι ότι ε, πρέπει να διατηρήσουμε τη διάκριση ανάμεσα στη μαύρη, στην γκρι και στην άσπρη λίστα ως προς την πρόσβαση σε αποδεικτικά έγγραφα. Και αυτό για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για να διευκολύνουμε τα αδύναμα μέρη και το δεύτερο να μην υπάρχουν αντιφάσεις από κράτος σε κράτος. Αυτό μεταφράζεται στην ψηφοφορία και κοιτάζω τον Ανδρέα ότι στις τροπολογίες που έχει καταθέσει είναι οι τροπολογίες από το 47, αριθμό 47 μέχρι το 61 ε, είναι τροπολογίες που ουσιαστικά αλλάζουν όλη την αρχιτεκτονική όλη τη στόχευση της οδηγίας. Mm. Αυτό σκεφτόμαστε. Και θέλουμε να το σκεφτεί και ο κύριος Βάπ. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε, όχι μόνο θέλουμε, οφείλουμε να υπερασπιστούμε το μαχητό τεκμήριο βλάβης σε περίπτωση παραβίασης του δικαίου του ανταγωνισμού. Το βάρος απόδειξης της βλάβης πρέπει λοιπόν κατά κατά τη γνώμη μας, να το φέρουν οι παραβάτες και όχι οι ζημιοθέντες. Και αυτό λόγω της ασυμμετρίας της πληροφόρησης που υπάρχει. Άρα αυτό μας οδηγεί στις τροπολογίες 87 και 89. Εδώ ε, τελειώνει το, το κομμάτι, το σύνολο των παρατηρήσεων, των επισημάνσεων που έχουμε να κάνουμε ως σοσιαλιστές, ως ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση. Και κλείνοντας, θέλω να και να υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η προσέγγιση του κυρίου Σμιτ ε, βρίσκει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα σημεία. Θα έλεγα ότι ε, η, η, προσέγγιση του κυρίου Σμιτ λειτουργεί ευεργετικά και τονίζω τη λέξη ευεργετικά για τους καταναλωτές, για τους Ευρωπαίους πολίτες σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη. Ε, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο δρόμος που τον ξεκίνησε, τον άνοιξε ο κύριος, ο κύριος Σμιτ κάνοντας ε, υπέρβαση, κάνοντας καινοτομώντας, ε, είναι ένας δρόμος που αν τον περπατήσουμε νομίζω ότι θα ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και αυτή την εμπιστοσύνη την έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πολύ μεγάλη ανάγκη για να μπορέσουν να ανταποδώσουν με τη δουλειά τους και πάλι υπέρ των καταναλωτών. Ε, η ψηφοφορία αύριο μας περιμένει και θέλω να πιστεύω και εγώ, όπως είπε και ο κύριος Βάμπ, ότι θα είναι μια ψηφοφορία που θα έχει θετικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Good. Uh, thank you very much. Um, I think Mrs. is next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 επιτυχία στις ε, διαπραγματεύσεις θα κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και να ψηφιστεί το εν λόγω έγγραφο κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ το εξής. Um, this is in the context of the that in my own country we're just Πρέπει να σας πω ότι εμείς στη χώρα μου προσπαθούμε επίσης να κάνουμε ε, αναθεώρηση της εθνικής μας ε, νομοθεσίας και προβλέπονται η προσθήκη κάποιων στοιχείων όπως ε, αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ. Ο συνάδελφος όμως κ. Θόρστη δεν πρέπει να πω ότι είναι και ιδιαίτερα ενθουσιώδης με την όλη συμβιβαστική πρόταση. Θα το συζητήσω το θέμα τον κύριο Σμιτ. περιπτώσει, γενικά πρέπει να πω ότι δεν βλέπω για ποιο λόγο οι συστάσεις της Επιτροπής ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν και τα δύο καθεστώτα opt-in και ε, opt-out να εφαρμοστούν συγχρόνως και όχι μόνο να επιλέγεται ένα. Πιστεύω ότι αυτό εξάλλου είναι κάτι το οποίο εμπίπτει σε περίπτωση αποζημιώσεων και στην εθνική νομοθεσία κάθε χώρας. Κάθε μία μπορεί να έχει τη δική της προσέγγιση λοιπόν η κάθε χώρα. Γι' αυτό σωστά εισαγάγει κατά την ε, απόψή μου η Κομισιό την ευελιξία. Επίσης, δεν μας ε, ενθουσιάζει ένα γενικότερο εγχειρίδιο εφαρμογής, αλλά ίσως κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Διότι πιστεύω ότι εκ των υστέρων και τα κάθε, κάθε εθνικό δικαστήριο είναι αυτό στο οποίο την διακριτική ευχέρεια ε, έγκυται και η εφαρμογή των αποφάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Όσον αφορά την τρίτη συμβιβαστική λύση. Εδώ προτείνει να συμπεριληφθεί και δική μου τροπολογία ο κύριος ε, ε, Σμιτ. Εγώ θα προτιμούσα όπως και ο κύριος Φαμπ ε, να το διαγράψουμε διότι κάπου έχει ε, συμπεριληφθεί. Και η τροπολογία 89 του κ. Σάρη είναι εντελώ διαφορετική από την ε, τροπολογία της Συμβαστική και εγώ δεν δέχομαι η δική μου να συμπεριληφθεί. Διότι εμείς είχαμε πει ακριβώς το αντίθετο. όσον αφορά την, ε, την ε, διαδικασία αυτή αποζημίωσης. Πιστεύω όμως ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με πνεύμα δικαιοσύνης και αυτό είναι κάτι το οποίο αποφασίζει κάθε χώρα μετά από τις ε, κατάλληλες έρευνες που γίνονται. Δεν δέχομαι λοιπόν αυτά τα οποία λέει ο κυρία Σμιτ, αλλά και κάποια καλά νέα για σας κύριε Σμιτ. Ε, είναι αποδεκτή από εμά η συμβαστική τροπολογία σας 4. Ελπίζω ότι θα σας ε, ικανοποιήσει αυτό που λέει το 4. Εν πάση περιπτώσει αυτές είναι οι απόψεις μας. Και καλή τύχη. Κύριε Σφάμπ, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος, ότι χρειαζόμαστε πραγματική πρόοδο και να προχωρήσουμε. Επίση, το θέμα των συλλογικών προσφυγών και το θέμα συνεργασία διασυνολικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το ζητάμε από την Επιτροπή, προσπαθούμε και πρέπει να βρούμε λύση ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη οι καταναλωτές όταν ε, υπάρχει ε, παραβίαση των κανόνων του σωστού ανταγωνισμού σε θέματα εμπορικών πρακτικών. Εάν δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κιούμπικ. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Uh, Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα κάνω σύντομο σχολιασμό. Όπως είπα και στην τελευταία συζήτηση για τις ε, συλλογικές προσφυγές. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ε, ε, καταναλωτές και είπαμε ότι η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι οριζόντια. Και όπως, όπως είπε ο Πρόεδρος, η σύσταση είναι αρκετά ευέλικτη που γίνεται γιατί θα πρέπει να έχουν περιθώριο ελιγμών τα κράτη-μέλη για να δουν πώς θα μπορέσουν όλο αυτό τον μηχανισμό να τον εφαρμόσουν και να μην περιοριστούν σε έναν μόνο μηχανισμό και προβλέπει η πρώτη συμβαστική τροπολογία. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε την σύσταση όπως προβλεπόταν θα δούμε σε δύο χρόνια ούτως ή άλλως σε ποιο μέτρο ε, θα ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη. Τώρα, για την μετακύληση, την περίφημη. Ε, και για τους έμεσους αγοραστές. Αυτά τα οποία λέγονται είναι σημαντικά, αλλά θα πρέπει να δούμε με κάποιο μηχανισμό πώς μπορούμε να αποτρέψουμε μια πολλαπλή, αν θέλετε, ε, ε, ευθύνη, αν θέλετε, αλλά θα δούμε. Τώρα, στην περίπτωση των καρτέλ, Ακούσαμε τι κύριο ο που πιστεύει ότι η χρησιμοποίηση των ε, τεκμηρίων και των αποδείξεων ίσως δεν είναι η καλύτερη διαδικασία. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει πάντα. Τι... Τα τεκμήρια είναι χρήσιμο πάντα και σε κάποιες περιπτώσεις ε, μας ε, βοηθά να καταλήξουμε σε αποτελέσματα. Αν δούμε ότι όντως όπως λέγεται το 95% των, ε, όπως αναφέρεται, των καρτέλ δημιουργούν πρόβλημα, όλη αυτή όλη διαδικασία, αυτή η τεκμήρια δεν νομίζω ότι είναι κακή. Εμείς απλώς θέλουμε να πούμε ότι όταν η ζημία, ότι πάντα όταν υπάρχει ζημία, ποτέ δεν είναι μηδενική. Εάν υπάρχει ζημία, το δικαστήριο και όλοι τα συμβαλώμενα μέρη θα πρέπει με τα κατάλληλα τεκμήρια να το αποδείξουν και να το εκτιμήσουν καταρχά. Και πιστεύω ότι μπορώ να σας πω τελειώνοντας ότι θα... Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστική λύση και θα μπορέσετε κι εσείς να περάσετε την έκθεση πριν από το τέλος της θητείας σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για όχι, για να ολοκληρώσει την ε, όλη συζήτηση. Δεν το λόγο και πάλι στον κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε καλή συνενετική λύση αύριο. Διότι ακούγοντά σας και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, μπορώ να προϋποθέσω ότι για κάποια θέματα Έχουμε καταλήξει συμφωνία. Και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή γνωμοδότηση στην ΕΚΟΝ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι ο κύριος Φόξ δεν ήταν και ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Δεν ζητούσα εγώ κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως. Απλώς στο, τέλος πατήσατε το σωστό κουμπάκι. Άρα κάναμε ένα βήμα προς τα μπρος. Διότι, εάν θέλουμε το όλο αυτό πρόβλημα να το ολοκληρώσουμε πριν από το τέλος της θητείας μας, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και όλος στόχος της υπαρξής μας εδώ, ξέρετε καλύτερα από όλους, ε, Πρόεδρε, εδώ είναι ότι πρέπει να φτάνουμε σε συμβιβαστικές λύσεις Είτε είμαστε πιο ικανοποιημένοι, λιγότερο ικανοποιημένοι. Πρέπει να το κατορθώνουμε κάποιον. Και στο τέλος η ECR πρέπει να σας πω ότι δεν θα μπλοκάρει μία συμβιβαστική λύση στην οποία θα καταλήξουμε. Διότι, ολοκληρώνοντας θα πω το εξή. δεδομένου ότι ασχολούμαι εγώ με τις ε, ασφάλειες, τις συντάξεις. Αν δούμε τι γίνεται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνησή σας ε, προσπαθεί να ρυθμίσει τα πάντα. Είναι εκπληκτικό τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση την δεξιά. Και εγώ που είμαι φιλελεύθερος πρέπει να πω ότι κάποια μέτρα τα οποία θέλετε να εισαγάγετε είναι θετικά, αλλά όχι και ιδιαίτερα φιλελεύθερα. Ίσως είναι φιλικά προς τον καταναλωτή, αλλά εν πάση ελπίζω ότι στο τέλος θα προσπαθήσετε <laughs> να έχετε μία πολύ μινιμαλιστική άποψη για να μπορέσουμε να καταλήξουμε αύριο στη συμβαστική λύση. Ευχαριστώ. <laughs> Σας ευχαριστώ για αυτή την προσεκτική ανάλυση του τι ακριβώς συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά πρέπει να σας πω επί τούτου ότι κάνουμε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση όσον αφορά τα θέματα προστασίας των κατανατών με την σύμπραξη των ενώσεων κατανατών και μας είναι ιδιαίτερα προσφυλέ τα θέμα αυτό των θέμητων πρακτικών. Ούτως ή άλλως, Νομίζω ότι θα υποστηριχθούν οι συμβαστικές λύσεις από πολύ μεγάλη πλειοψηφία και μετά το μπαλάκι θα περάσει στον κύριο Σφάμπ. Πολύ καλά. Τώρα βλέπω ότι είναι 5.30, έχουμε μια τελευταία έκθεση. Βλέπω ότι τώρα μόλις φτάνει ο εισηγητής, θα τον περιμένω να καθίσει για να μας παρουσιάσει το επόμενο θέμα του. Το πακέτο που αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες οργάνωσης ταξιδίων. Ακούσαμε σε ακρόαση τους εμπειρογνώμενους, έκανε έκθεση την οποία μας παρουσίασε ο κύριος Μάιερ, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών την πέμπτη αυτή τη εβδομάδα. Νομίζω ότι το ξέρατε όλοι και ήδη έχουν τέτοιο τροπολογίες και τώρα θα του δώσω τον λόγο αλλά πριν ο κύριος Κοφεράτη ο αντιπρόεδρος μας είναι εδώ δεν ξέρω αν έρθει κάποιος εκ μέρους των φιλελευθέρων. Α, σκιώδης ο κύριος Σμιτ για αυτό το θέμα. Η κυρία Ρούρε είναι σκιώδη σε όλα τα θέματα σήμερα το απόγευμα. Κύριος Τεγιόν και ο κύριε Σαγκίνη δεν είναι εδώ. Είναι εδώ κάποιος από την Κομισιόν. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι. Η κυρία Μανφρέντι από την Κομισιό. Και ο κύριος Ματιάκ. Χαίρομαι που σας βλέπω και τους δύο εδώ. Σήμερα το απόγευμα. Ας αρχίσουμε τη συζήτηση. Δίνω πρώτα απ' όλα το λόγο στον κύριο Hans Peter Mayer. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας για τη συζήτηση αυτού του θέματος και σας υπενθυμίζω ότι το κοκτέιλ θα αρχίσει ακριβώς στις 6. Όσο λοιπόν περισσότερη ώρα περάσουμε εδώ, τόσο λιγότερο χρόνο θα έχουμε για τα ποτάκια μας. Ο εισηγητής πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε με πολύ χαρά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτού ασχοληθώ με την ουσία της εισήγησής μου. Ήταν πάρα πολύ ε, δύσκολο να λάβω υπόψη όλες τις θέσεις διότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε με όλους και να καταλήξουμε σε μια ισορροπία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο αλλά είμαι ε, πεπισμένος ότι δεν θα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Είμαι πάντοτε ανοιχτός για περαιτέρω συζητήσεις κυρίως για τις ε, τροπολογίες που θα κατατεθούν από τους συναδέλφους και εγώ προσωπικά θα προτείνω ορισμένες βελτιώσεις ε, σε σχέση με τα όσα έχω πει. Ε, ξέχασαν οι μεταφραστές να μεταφράσουν την τροπολογία υπαριθμών 1, διότι νόμιζαν ότι είναι ένα, πρόγραμμα, ένα πρόβλημα γλωσσικό, αλλά είναι ένα πρόβλημα ορισμού. Πρόκειται για την ίδια την αντίληψη linked travel arrangements, εξατομικευμένες υπηρεσίες πρέπει να δούμε αν μια εναρμόνιση ελάχιστη ή μέγιστη πρέπει να επιτευχθεί. Η θέση της Κομισιόν δεν είναι σαφής. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν παρόμοια προστασία και δικαιώματα σαφώς καθορισμένα. Δεν θα πρέπει και από τις δύο πλευρές των συνόρων να αλλάζουν οι κανόνες θα πρέπει να έχουμε μία μόνο εσωτερική αγορά και αυτό έχει σχέση με την προστασία των καταναλωτών για να το εξασφαλίσουμε αυτό. Έλαβα υπόψη την διατύπωση της οδηγίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών που υιοθετήθηκε πριν από λίγο καιρό και που δεν ήταν πολύ επίμαχη και εκεί λέει ότι στο σημείο όπου η οδηγία ισχύει, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να έχουν προδιαγραφές που να διείστανται από το κείμενο αυτής της οδηγίας. Και αυτό για... ισχύει για τους κανόνες που θα επέφεραν μια άλλου είδους προστασία. Για την προστασία λοιπόν των καταναλωτών θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε πάντοτε τους ίδιους κανόνες, ταυτόσιμους κανόνες. Δεν θέλω να μειώσω την ποιότητα της προστασίας των καταναλωτών. Θέλουμε μια καλή προστασία των καταναλωτών και θα πρέπει να επιτύχουμε να θεσπίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας παντού. Βεβαίως μπορούμε να προβλέψουμε εξαιρέσεις στον κανόνα, μπορούμε στον νόμο να προβλέψουμε εξαιρέσεις, παραδείγματος χάρη οι Γερμανοί μπορούν να χρησιμοποιούν ε, μια πιο προχωρημένη προστασία των καταναλωτών, η Γαλλία θα επιθυμούσε επίσης μια προστασία για τις, ε, τους πράκτορες ταξιδιών, ε, για τους ενδιαμέσους δηλαδή, τους μεσολαβητές, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται είναι οι λέσχες, τα πανεπιστήμια, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις που οργανώνουν και αυτές ταξίδια, αλλά δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του κειμένου αυτού. Και συνεπώς η διατύπωση που προτάθηκε από την Κομισιόν αντικαταστάθηκε από την διατύπωση που εγώ πρότεινα στην τροπολογία μου σχετικά με τα επαγγελματικά ταξίδια και τα επιχειρηματικά. Αν μπορεί να υπάρξει ένα συμβόλαιο πλαίσιο, δεν θα πρέπει η επιχείρηση να είναι εξειδικευμένη στην οργάνωση των ταξιδιών, αλλά αν μια επιχείρηση έχει ένα συμβόλαιο πλαίσιο και οργανώνει τακτικά ταξίδια, και πάλι αυτό δεν πρέπει να ισχύει. Ε, στο άρθρο 2 συμπλήρωσα επίσης το κείμενο και είπα ότι οι παροχές που είναι απλώς παροχές δευτερεύουσες, συμπληρωματικές ε, στις βασικές δεν θα έπρεπε να αποτελούν ένα ταξίδι. Παραδείγματο χάρη ένα πρακτορείο ταξιδίων, ένα γραφείο ταξιδίων που έχει συνάψει ένα συμβόλαιο και που οργανώνει μόνο την μεταφορά προς το αεροδρόμιο, δεν πρέπει να, να θεωρηθεί αυτό συμβόλαιο ξεχωριστό, εφόσον είναι μέρος του πλαισίου των άλλων παραχών. Και δεν είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός να το αντιμετωπίσουμε. Δύο συμπληρωματικές δευτερεύουσες παροχές δεν πρέπει να καλύπτονται στο πεδίο εφαρμογής, παραδείγματος χάρη. Απλώς ένα ταξίδι με ε, νυχτερινό τρένο, με κουκέτες ή κρατήσεις. Δεν πρόκειται τότε ε, για ένα ε, ταξίδι πακέτο με μια μοναδική τιμή, με μια συνολική τιμή και για τα ξενοδοχεία ε, δεν πρέπει να ασκήσουμε πολύ πίεση. Οι απλές διανυκτερεύσεις ξενοδοχείου με διευθετήσεις που δεν είναι το βασικό στοιχείο αλλά δευτερεύον στοιχείο δεν θα έπρεπε να καλύπτονται από το κείμενο αυτό. Αλλά αυτό που είναι διαφορετικό είναι η περίπτωση όπου αυτό αποτελεί την βασική παροχή, τη βασική υπηρεσία. Θέλω να περάσω ε, να πάω κάπου σε μια συνάντηση και θα πρέπει να κάνω μια διενεκτέρευση επιτόπου. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο του ταξιδιού, τι προσδιορίζει το ταξίδι. Και εδώ μπορείτε να δείτε τις ε, προτάσεις που έχω κάνει. Άλλο σημείο έχω αυτό το ε, του Μπόλστάιν Ράιζε, τη βασική αντίληψη ε, που την άλλαξα σε οργανωμένο ταξίδι. Η πληροφόρηση πριν από τη σύναψη του συμβολέου. Εδώ δεν πρέπει να δίνουμε πολλές πληροφορίες στον καταναλωτή, διότι αυτό δεν γίνεται πολύ σαφές και διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην βλέπουμε τα βασικά στοιχεία της προστασίας του καταναλωτή. Είναι η δυνατότητα να μπορούμε να αποσυρθούμε, να έχουμε τη δυνατότητα να ακυρώσουμε κλπ. Το πέμπτο σημείο είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου λείπει από την πρόταση της Κομισιό, είναι η δυνατότητα ακύρωση συμβολέων θα πρέπει ο ταξιδιώτης να μπορεί να αποσυρθεί, να έχει μια προθεσμία 24 ώρες αλλά αυτό δεν ισχύει για τα συμβόλαια ε, που συνάπτονται την τελευταία στιγμή, δηλαδή λιγότερο από 15 μέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης να εισαχθεί για την προστασία των καταναλωτών, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν πάντοτε την δυνατότητα να αποσυρθούν, να ακυρώσουν, εάν παραδείγματος χάρη το ταξίδι καθίσταται ανέφικτο λόγω ανωτέρας βίας, πολέμου, ασθένειας κλπ. Θα πρέπει να μπορεί να ακυρώσει το συμβόλαιο χωρίς έξοδα. Αλλά αυτό να μην είναι εφικτό εάν ο ταξιδιώτης ήξερε εκ των προτέρων αυτά τα στοιχεία όταν κράτησε το ταξίδι και δεν τα έλαβε υπόψη. Νομίζω ότι τότε είναι δική του ευθύνη. Έκτο σημείο στο μέτρο όπου υπάρχει αλλαγή ταξιδιού από τον οργανωτή και είναι κάτι σημαντικό θα πρέπει ο ταξιδιώτης να έχει τη δυνατότητα κύρωσης του συμβολέου χωρίς να έχει να υποστεί συνέπειες συμπληρωματά Θα, μπορεί, θα πρέπει να μπορεί να ακυρώσει όλο το ταξίδι. Θα πρέπει τότε να είναι εξασφαλισμένος να έχει κάποια ασφάλεια για τις διακύμανσεις τιμών. Αυτό ισχύει ε, για τα ταξίδια που έχουν κρατηθεί πριν από πάρα πολύ καιρό. Αν υπάρχει μια αύξηση τιμής, δεν θα πρέπει να μετακυλιστεί ε, στον καταναλωτή αν είναι πάνω από ε, αν είναι μόνο αν είναι πάνω από 3%. Αν είναι πολύ μικρή δεν θα πρέπει να μετακυλίεται να επιβαρύνει τον ταξιδιώτα είναι λιγότερο από 3%. Δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά μια μείωση τιμών θα πρέπει να ισχύει αν είναι προς όφελος του καταναλωτή. Και εδώ λοιπόν έχουμε εισαγάγει αυτό το 3% αλλά εφόσον υπάρχουν πάντοτε διοικητικά έξοδα θα πρέπει να μπορούμε να προβλέψουμε ένα ποσό που σε κάθε περίπτωση θα μπορεί να εισπραχθεί από το γραφείο ταξιδίων και αυτό είναι κάτι στο όν υπάρχει μια αύξηση τιμής άνω του 10% αυτό αποτελεί σημαντική αλλαγή του συμβολέου και αυτό θα έπρεπε αυτομάτως να δίνει την δυνατότητα ακύρωσης ή την δυνατότητα να του προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι δύο τύπου για την τιμή, την αρχική τιμή. Πολύ συχνά έχουμε την τάση ε, να το βλέπουμε αυτό πολύ αργά, βάζοντας χάρη ένα ταξίδι για τέσσερα άτομα, κανείς πρέπει να πληρώσει 10% επιπλέον, αυτό είναι σημαντικό εμπόδιο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Σε μια τέτοια περίπτωση το γεγονός ότι απλώς έχει κανείς ε, την δυνατότητα ακύρωσης θα πρέπει να την έχει. Ε, και δεν αρκεί αυτό, διότι θα πρέπει η οικογένεια να βρει μια άλλη δυνατότητα και σε εποχή εχμής θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν το γραφείο του ταξιδίου να του κάνει μια εναλλακτική ε, λύση. Θα πρέπει να έχει να διαλέξει ανάμεσα σε τρεις επιλογές αν υπάρχει αύξηση άνω του 10% μπορεί να δεχθεί ε, βεβαίω το ταξίδι με την ευξημένη τιμή, να δεχθεί ένα άλλο ταξίδι που θα προτεθεί, η τρίτη δυνατότητα να ακυρώσει το ταξίδι με επιστροφή του ποσού που έχει ήδη καταβάλει. Μετά έχουμε την προστασία κατά της αφαιρεγγιότητας. Αυτό ισχύει όχι μόνο από οικονομικής απόψεως για την ανάκτηση των χρημάτων, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι δεν θέλουμε πάντοτε ε, να ε, να τα πάρουμε όλα. Ε, μπορεί να θέλει ο ταξιδιώτης να συνεχίσει το ταξίδι. πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών στην περίπτωση όπου έχουν κρατήσει ένα τέτοιο οργανωμένο πακέτο ταξιδιού. Όσον αφορά στην ευθύνη, Νομίζω ότι στην περίπτωση όπου δεν μπορεί κανείς να επιστρέψει τα χρήματα λόγω ειδικών συνθήκων, τότε ο οργανωτής είναι υπεύθυνος και θα πρέπει πάντοτε να προβλέπει τουλάχιστον μια εναλλακτική λύση για τους ταξιδιώτες. αν είναι σαφές ότι ο οργανωτής δεν μπορεί δεν επιθυμεί να το πράξει, αυτή είναι η περίπτωση όπου έχουμε την υποχρέωση να προβλεφθεί μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο για τον ταξιδιώτη σε περίπτωση όπου ακινητοποιηθεί. Η πρότασή μου προβλέπει ότι ο ταξιδιώτης που θα πρέπει μόνος του να αναζητήσει ξενοδοχείο Μπορεί ε, για λίγες μέρες χωρίς όριο και πάνω από πέντε μέρες με όριο που προβλέπεται από την Επιτροπή. Έλαβα πολλές διαφορετικές ιδέες και εδώ δεν είπαμε την τελευταία μας λέξη και δεν λήφθηκε η απόφαση. Αύριο είναι η Επιτροπή Μεταφορών που θα αποφανθεί για το θέμα αυτό και θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Στην περίπτωση όπου υπάρχει μια μείωση τιμής, εγώ είμαι της γνώμης ότι ότι δεν είναι μόνο ο ταξιδιώτης που θα πρέπει να αναλάβει τον κίνδυνο, αν υπάρχει ο κίνδυνος, ο κίνδυνος θα πρέπει να μοιραστεί 50-50 ανάμεσα στον ταξιδιώτη και στο γραφείο ταξιδίων, διότι ούτε το γραφείο ταξιδίων, ούτε ο ταξιδιώτης δεν πρέπει να θεωρηθεί πλήρως υπεύθυνο για... Kürzere gewählt. Vielen Dank. Έδωσα μια γενική εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις διεξοδικές σας παρατηρήσεις. Έχουμε και χρόνο στην ε, διάθεσή μας να ακούσουμε τώρα τους σκιώδες εισηγητές για τις δικές τους συνεισφορές. Ο κύριος Κοφεράτη να ξεκινήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σημαντικό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει αυτή την οδηγία, διότι έρχεται να καλύψει Κάτι που με την πρώτα του χρόνου δημιουργήθηκε, ένα κενό δηλαδή, ένα διαρκές κενό που φαινόταν ότι υπήρχε σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Να θυμηθούμε την οδηγία του 90 που ήταν η προηγούμενη και το πόσο άλλαξε με το χρόνο αυτή η δραστηριότητα ακόμη και με την τόσο ευρεία χρήση του διαδικτύου και των, πληροφοριακών, των πληροφορικών δυνατοτήτων. Αυτό το κενό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Ο χρόνος που πέρασε επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον εισηγητή να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από νέα επιχειρήματα, όπως είδαμε και από τις προτάσεις που μας ε, παρουσίασε μόλις τώρα ο εισηγητής. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, για λόγους οικονομίας του χρόνου και δεν θέλω να μπω σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Θέλω να εμείνω σε, μερικές μόνο, σε μερικά μόνο σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά για τη λειτουργία της Επιτροπής μας. Εμείς ασχολούμαστε κατεξοχήν με τους καταναλωτές. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε έτσι ώστε όλες οι προδιαγραφές για το θέμα αυτό να διαπανταπονομική ασφάλεια και να είναι και εύληπτες όπως είπε και ο εισηγητής. Αυτό θα πρέπει να είναι η, το σημείο αφετηρίας. Βεβαίως και για τις υλικέ συνέπειες, για όσους διέπονται από τους κανόνες για τους οποίους συζητούμε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πάντως κάποιες πτυχές πρέπει να εξεταστούν. Είναι αντικειμενικά πιο σημαντικές από άλλες. Δεν θέλω να υποτιμήσω κάποιες από τις παρατηρήσεις ή τις λεπτομερείς, ε, ε, τα λεπτομερή σχόλια που θα κάνετε, αλλά στις, στην καθημερινότητα κάποιες συμπεριφορές πρέπει να προστατεύονται κατά προτεραιότητα. Λόγου χάρη, αν υπάρχει μια σοβαρή αλλαγή στον ορισμό της τιμής ενός πακέτου Αναγκαίο θα είναι να υπάρξει και ρητή συνένεση από την πλευρά του καταναλωτή. Ξέρουμε ότι σήμερα αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Οι αλλαγές που οφείλονται σε οποιοδήποτε αίτιο στην καθημερινή πράξη πολλές φορές αντιμετωπίζονται με σχετική συνέπεια. Πριν λοιπόν οριστεί νέα τιμή για ένα πακέτο, καλό θα είναι και σημαντικό είναι ο καταναλωτής να γνωρίζει και ρητός να συγκατατίθεται. Έπειτα η Επιτροπή προβλέπει ένα όριο για την αύξηση της τιμής. Είτε σου φορά την ίδια την αύξηση είτε και τον χρόνο ενημέρωσης. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ συχνό φαινόμενο. και έτσι εκδηθετεί καταναλωτέ σε κινδύνου. Θεωρώ και σημαντικό και αναγκαίο να περιοριστεί αντιπεραιτέρω η δυνατότητα και κατά συνέπεια η ευχέρεια του, παρέχοντα να αυξήσει την τιμή και του ορίου που ε, προβλέπει η Επιτροπή, να μην βρεθεί στην δύσκολη θέση ο καταναλωτή να μην μπορεί να διαλέξει, να υπάρχουν και εναλλακτικέ. Δηλαδή τι εννοώ, εάν υπάρχουν θεωρητικέ εναλλακτικέ, δεν αρκεί, διότι τελικά δεν εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη επιλογή. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα που δεν νομίζω ότι κατά τύχη μα σχολίασε ο εισηγητή με μια σειρά από υποθετικά σενάρια, τα οποία καλό θα είναι να τα σκεφτούμε, της πλήρους ενημέρωσης, της ε, ενημέρωσης με σκοπό την πρόληψη. Το περιεχόμενο όμω τη ενημέρωση αυτή καθεαυτή, αλλά και το πώ χρησιμοποιούνται οι πληροφορίε οι οποίε παρέχονται, αυτό είναι σημαντικό. Διότι ξέρουμε ότι είναι πολύ διαφορετικέ οι συμπεριφορέ των καταναλωτών μεταξύ του. Υπάρχουν καταναλωτέ που έχουν καλή σχέση με τα εργαλεία τη πληροφορική και άλλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνο τα έντυπα και μόνο σε αυτά βασίζονται. Το είδος λοιπόν, ο χαρακτήρας της πληροφορίας αλλά και τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να μπορούν να επιλέγονται κάθε φορά αναπερίπτωση από τον καταναλωτή, ώστε όσοι ταξιδεύουν να μπορούν να ταξιδεύουν σε συνθήκες ασφάλειας, με, τη μέγιστη, με το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας. Ιδίω σε ό,τι αφορά αυτή τη διάσταση της ενημέρωσης, μπορούμε να εμπνευστούμε από τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε στην Επιτροπή μας και για ένα άλλο θέμα, τελείως διαφορετικό. Όταν συζητήσαμε την ενημέρωση κλειδί για τις επενδύσεις. Εδώ δεν μιλούσαμε για μεμονωμένους καταναλωτές, αλλά για την επιχειρηματική διάσταση, τις εταιρείε, οι οποίες ε, συνηθίζουν και είναι εξοικειωμένες με αυτό το είδος της πρακτικές. Εκεί έγινε επιλογή και διάκριση πολύ ακριβής, πολύ προσεκτική, όπου κατά τη γνώμη μου ε, εμπεριείχε ένα κριτήριο το οποίο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε μετατρέποντάς το και σε ε, όρο, προϋπόθεση που να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και του εισηγητή θα πρέπει σε όσους εκπροσωπούμε να τους δώσουμε την ε, βεβαιότητα ότι εμείς στο διάστημα αυτό από το 1990 ως σήμερα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι εύστοχο. Και ότι δεν υπήρχαν αρνητικές προθέσεις στο κατά πόσο καλύπτονται, αλλά στο ότι άλλαξαν πάρα πολύ τα πράγματα, το σκηνικό γύρω μας. 25 χρόνια σχεδόν ε, οι κανόνες του παρελθόντος δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παρόντος, είναι απαρχιωμένοι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Thank Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω εδώ μια δήλωση. Εκ μέρους του κυρίου Χατζημαρκάκη. Ευχαριστεί τον εισηγητή για την επιμελή του εργασία του φακέλου αυτού και την επιδίωξη του να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των κατώμελών. Καθώς η Ευρώπη είναι ο πλέον προσφυλής τουριστικός προορισμός, είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε κοινού επικαιροποιημένους νόμους που να διέπουν τις επιλογές και τις διαδικασίες τις βάλλονται οι ταξιδιώτες. Ο κ. Χατζημαρκάκης αναγνωρίζει την ανάγκη να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες, οι καταναλωτές τι αγοράζουν και βεβαίω και του ε, κανόνε περί αφαγγελέτα και το καθεξή. Θέλει να τονίσει ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε τι τοπικέ επικοινωνίε που μπορεί να πληγούν εάν δεν προβλεφθούν δυνατότητες και για μικρότερες εταιρείες που λειτουργούν τοπικά από το πακέτο για την προστασία των ταξιδιωτών, όπως επίσης να μην είναι παράλογα τα ποσά της αποζημίωσης. Πρέπει να είναι ε, ανάλογα με το ποσό του πακέτου που αγοράζεται. Τώρα εγώ προσωπικώς θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Μάγερ. Προτείνεται πλήρη εναρμόνιση εδώ. Πλήρη εναρμόνιση και στο κείμενο αναφέρεται δύο πόλεις, το Άχεν και άλλη μια πόλη που αποθέτωται βρίσκεται στα σύνορα με την Ολλανδία. Α, στο Βέλγιο είναι. Ωραία, εντάξει. Τέλο πάντων, είναι δύο πόλει ε, κοντά στα σύνορα Ολλανδία-Βελγίου. Ήθελα τα σχόλιά σα εδώ. Είναι εφικτό αυτό. Μπορεί να γίνει. Η πλήρη μέγιστη δυνατή ενερμόνιση, Γιατί αυτό προτείνεται. Καταλαβαίνετε, είναι κάπω περίπλοκο. Και η άλλη με ερώτηση είναι η εξή. Όλοι εμείς ταξιδεύουμε. Με πακέτα και χωρί. Πού είναι το όριο της ευθύνης. Το όριο της προσωπικής ευθύνης του καθενός. Διότι έχω την αίσθηση ότι το όριο αυτό όλο ένα και μειώνεται, κατεβαίνει. Είναι λες και το άτομο που ταξιδεύει δεν έχει την ευθύνη του αυτού του. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε λίγα και αυτό, αν μπορείτε να το αναπτύξετε, διότι καταστροφές υπήρξαν και υπάρχει πάντοτε η εντύπωση ότι αν κάτι πάει στραβά δεν προστατευόμαστε και ούτε κυβέρνηση θα μας σώσει. Καταλαβαίνω τα επιχειρηματά σα, αλλά θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα ε, τη σήμερα ημέρα. Ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ κύριε Αρούλε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Νομίζω ότι έκανε πολλή δουλειά σε πολύ λίγο χρόνο. Και έχει διευκρινίσει πολλά στοιχεία που ήταν πολύ συγκεκριμένα τώρα. Όμω ακόμη παραμένουν να κρεμίσει κάποιε ερωτήσεις. Έχω και εγώ την ίδια ερώτηση με τον κύριο Σμιτ. Και εγώ διερωτώ με εάν μπορούμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αρμόνιση. Δεν υπάρχουν άλλοι τομεί στου οποίου θα έπρεπε να γίνεται αυτή τόσο μεγάλη προσπάθεια. Στον τουρισμό θα επιμείνουμε. Να προσαρμοστούμε, δεν λέω, αλλά τέτοια πίεση για την προσαρμογή στι αλλαγέ την αντιμετωπίζουμε διαρκώ τα τελευταία χρόνια, μόνο και μόνο με την ύπαρξη του διαδικτύου. Οπότε, διερωτώ με, η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση είναι ό,τι καλύτερο. Πόσο θα πιέσουμε τα κρατημέλη. Δεν είμαι πεπισμένη. Ό,τι είμαι πεπισμένη ότι έχουμε βρει τη βέλτιστη λύση για το πεδίο εφαρμογής. Εγώ πάντοτε αντιμετωπίζω δυσκολίες με το θέμα των οργανωμένων ταξιδιών με τα πακέτα, τα ταξιδιωτικά και όλα τα σχετικά στοιχεία. Εδώ υπάρχουν τομεί που επικαλύπτονται. Τομεί όπου υπάρχουν, υπάρχει προσφορά υπηρεσιών και που θα εκλείψουν εάν αρχίσει να συνδέεται όλο αυτό με τα προστασίας ή και πτωχεύσει ε, εάν αρχίσουμε να συζητάμε με τέτοια μονή τη αποζημιώσεω και το καθεξής. Δεν είναι πάντως όλα σαφή και όπως είπατε κύριε Σμιτ, Τι εννοείται κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι πλήρης, δεν αρκεί να είναι διαφανής. Να ξέρει ο καταναλωτής τι κίνδυνο αναλαμβάνει, αλλά αυτό δεν φτάνει. Τρίτη παρατήρηση. Το θέμα των επαγγελματικών ε, μετακινήσεων και ταξιδιών. Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως ξεχωριστή κατηγορία. Δεν είναι διαφορετικό από τους μεμονωμένους ταξιδιώτες. Θα έπρεπε να καλύπτεται και αυτό από αυτή την οδηγία. Νομίζω εδώ θα χρειαζόταν μια γενική εξαίρεση για τα επαγγελματικά ταξίδια. Πάντως, ομολογώ ότι έχω εντυπωσιαστεί όπω θα κάνατε σε τόσο λίγο χρόνο, κύριο Μάγερ, και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να συζητούμε ε, επικοδομητικά. Αυτά από τους άντρους, κυρία Μακλάρκη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με σκέφτεσαι εισηγείται για το θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι πρόκειται για ένα τμήμα του δικαίου που πρέπει όντω να επικαιροποιηθεί. Όχι μόνο στα πλαίσια τη σύγχρονη αγορά, αλλά γιατί πραγματικά χρειάζεται ένα επιπλέον επίπεδο σαφήνεια για του καταναλωτέ, του ε, ταξιδιώτε και να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά του και τι καλύπτεται. Επ' αυτόν όμω θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς εξετάζουμε, πώς μπορούν να κάνουν καλύτερες επιλογές οι καταναλωτές χάρη στην ενημέρωση που λαμβάνουν, αλλά μην αφαιρέσουμε και τη δυνατότητα δράσης των επιχειρήσεων, ούτε να δυσκολέψουμε και τους καταναλωτές, να με βρίσκουν περισσότερες, πολλές προσφορές δηλαδή. Να εργαστούμε λοιπόν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά μην ξεχνάμε και τι επιχειρηματικέ ανάγκε. Τα συζητάγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθούμε σε κάποιου τομεί, να του συζητήσουμε σε αυτή τη φάση και μετά για ένα μεταγενέστερο στάδιο να αφήσουμε κάποια άλλα στοιχεία. Πάντω οι καταναλωτέ θα πρέπει να είναι βασικοί δικαιούχοι, του οποίου αφορά αυτή η πρόταση και είναι και περισσότεροι. Ε, πελάτε θα πρέπει να εξαιρεθούν εδώ οι επιχειρήσει. Έχουμε μια τροπολογία σχετικά για του επαγγελματίε ταξιδιώτε, για τα επαγγελματικά ταξίδια οι οποίοι θα πρέπει να το επισημαίνουν αυτό τη στιγμή της κράτησης και αυτό διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά να επικεντρωθούμε όντως στις περιπτώσεις των αναμονωμένων ταξιδιωτών, διότι οι επιχειρήσεις διαφέρουν. Έχω πρόβλημα με τον όρο assisted travel, εξατομικευμένες υπηρεσίες. Εδώ θα πρέπει αυτό κάπως να μετονομαστεί σε linked travel, συνδεόμενη υπηρεσία. Διότι δίνεται η εντύπωση ότι κάποιος ε, ε, δράος μεσάζων για να προσφέρει μια υπηρεσία που έχει σχέση με το ταξίδι. Όχι, το linked είναι ίσως ο καλύτερος όρος για να το ορίσουμε αυτό, να το διευκρινίσουμε. Τη στιγμή που θα κοιτάμε τους ορισμούς, νομίζω θα δυσκολευτούμε περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της πρότασης με αυτό, γιατί πρέπει εμεί οι ίδιοι να κατανοήσουμε τι εννοούμε με του ορισμού, το ίδιο και στις επιχειρήσει, αλλά στο τέλο πρέπει να καταλαβαίνουν και οι καταναλωτέ τι καλύπτεται και τι όχι και ποιε είναι οι υποχρεώσει και τα δικαιώματά του. Και ο κλάδο επίση των επιχειρήσεων θα θέλει να ξέρει πώ θα ενημερώνονται οι καταναλωτέ. Πρέπει και εμεί να το καταλάβουμε για να βρούμε ένα πραγματικά αποτελεσματικό τρόπο να φτάνουν οι πληροφορίε εκεί που πρέπει. Επίση, με απασχολεί τι θα γίνει με τον ορισμό του σημαντικού μέρου του πακέτου των προσφορεμένων υπηρεσιών. Το 20% αναφέρεται εδώ ω ποσοστό για ένα πακέτο και αυτό θεωρείται ένα σημαντικό ποσοστό. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα το δουν έτσι και οι καταναλωτέ. Το 20% θα το βρουν σημαντικό, σοβαρό ποσό ή όχι. Πρέπει να δούμε πώ οι επιχειρήσεις πολλούν τα πακέτα αυτά προ του καταναλωτέ. Εάν συμπεριλαμβάνουν και άλλε υπηρεσίε πέραν του ταξιδιού, θα πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη και να σκεφτούμε πώς αυτό το ποσοστό αλλάξει, μήπω η ζυγαριά κλείνει προ την άλλη πλευρά. Μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή μια βοηθητική υπηρεσία, γιατί αυτό θα είναι δύσκολο να οριστεί από την πλευρά του καταναλωτή να, το κατανοήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για την ε, εξάλληψη της υποχρεωτικής εκτύπωσης. Εγώ δεν θέλω να συνεχίσουμε να προσθέτουμε άχθη στι επιχειρήσει, γι' αυτό υπέβαλα τέτοιε τροπολογίε για την ε, ενημέρωση των ε, πληροφοριών σε σχέση με τι διακοπέ. Αυτό που περισσότερο αλλά πραγματικά με απασχολεί και η εναρμόνιση των ε, ε, συμβάσεων του καταναλωτικού δικαίου. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό και κάποια κάτι μέλη ήδη χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται ωφέλη που από αλλού. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν θα επιτρέψουμε στα κάτι μέλη να εφαρμόσουν ή να επιτρέπουν την ισχύ των αυστηρότερων ε, διατάξεων εφόσον ήδη τις προβλέπουν στην νομοθεσία τους. Νομίζω τα ταξιδιωτικά πακέτα και οι συνδεόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να διακριθούν από τα, σε δύο κατηγορίες από τα, τα τα πούλμαν από τις αεροπορικές ε, μετακινήσεις. θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη η στόχευση της κάθε διάταξης, διότι δεν θα είναι σαφής η νομοθετική μας πρόταση για το τι είδους υπηρεσία παρέχεται και για τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται. Το πώς θα διαφοροποιήσουμε τώρα τα πακέτα. Και αν θα μιλάμε για εξατομικευμένες συνδυόμενες υπηρεσίες, πώς θα το κάνουμε αυτό όταν μιλάμε για ένα σύνολο, ένα πακέτο που κλείνει κανείς για μια στιγμή δηλαδή. Αυτό θα είναι το πακέτο και τα συνδεόμενα θα είναι αυτά που τα κλείνει κανείς το ένα μετά το άλλο μέσα σε ένα 24ωρο. Μήπως παίζει ρόλο το χρονικό περιθώριο. Ή το δικαίωμα απόσυρσης επίσης. Άρνησης. Οι διακοπές της τελευταίας στιγμής. Οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής. Θα είναι πολύ δύσκολο αυτό να προσφέρεται Διότι μπορεί να το αγοράζει αυτό ο καταναλωτή, αλλά πώ θα συμπίπτει αυτό με το χρόνο άρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε ακριβώ αυτό, του ορισμού σε σχέση με το δικαίωμα άρνηση. Πάντω, ε, μπράβο σα για τη δουλειά σα ω τώρα, γιατί έχει πολύ ακόμα δουλειά να γίνει η πρόταση αυτή για να είναι έτοιμη, αλλά θα χρειαστούν εντατικέ συνομιλίε για να βρούμε λύσει σκεπτόμενοι, σκεπτόμενοι το τι θα γίνει με τους καταναλωτές βέβαια και τις ανάγκες τους αλλά και με τις επιχειρήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έχω ακόμα τρεις συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν, η κυρία Στάιλερ, η κυρία Χάνσλι και η κυρία Βάιλερ. Μπορείτε να κάνετε και εσείς τα σχόλιά σας, αλλά θα ήθελα και λίγο χρόνο για να ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη γιατί βλέπω ότι μας πιέζει ο χρόνος και εγώ Συνολικά καλωσορίζω την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα όσα κάνει ο εισηγητής. Κύριε Μακλάκιν, μίλησε για το assisted travel. Στα αγγλικά κιόλα υπάρχει πρόβλημα με τις εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ίσως τη στιγμή που θα μελετήσουμε τους ορισμούς θα πρέπει να το σκεφτούμε καλύτερα. Linked, συνδεόμενες ίσως είναι πολύ καλό να το πούμε. Εγώ Όταν ε, άρχισα να δουλεύω, ήμουν βοηθός ε, βουλευτού στο ε, Βρετανικό Κοινοβούλιο και κάποιες φορέ, επειδή ήμουν ακριβώ βοηθό και συνόδευα τη βουλευτή σε κάποια ταξίδια τη, μιλούσαμε για assisted travel, για, για ταξίδι όπου υπήρχε συνοδεία, διάσταση συνοδεία. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο κάποιο είδου ταξίδια που κάποιο συμμετέχει ω επιπλέον μέλο Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ περιπτώσει λοιπόν. Είναι πολύ καλύτερα να μιλάμε για link, για συνδεόμενε υπηρεσίε, παρά για τόσο συγκεκριμένε ή ειδικέ κατηγορίε που ήδη έχουν κάποιο άλλο νόημα. Επίση, θα πρέπει να προσέξουμε να μην είναι πολύ στενό ή περιορισμένο το πεδίο τη οδηγία, το κατά πόσον θα δημιουργήσουμε άγχο για τι μικρότερε επιχειρήσει, αλλά όταν να υπάρξουν και παραθυράκια δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα δημιουργήσει καινούργια παραθυράκια σε σχέση με αυτά που υπάρχουν. Θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε το σωστό και αυτό είναι σημαντικό από την πλευρά τη προστασία των καταναλωτών. Επίση, το είπε και ο κύριο Κοφεράτη, θα πρέπει να είμαστε σαφεί και ε, εύληπτοι στι ε, πληροφορίε που θα δίνουμε. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε σωστά ε, την ιεράρχηση των αναγκών που θέλουμε να καλύπτουμε. Ευχαριστώ πάντω τον εισηγητή, ευχαριστώ και του Σκιώδη και ε, νομίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι την Τετάρτη. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά ελπίζω να το ξανασυζητήσουμε, Πρόεδρε, όλοι μαζί από τον καινούργιο χρόνο. Ευχαριστούμε, κυρία Χάνσλικ. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συνάδελφο. Συμφωνώ με την πλειοψηφία των υποδείξεων και παρατηρήσεων που έκανε ο εισηγητής. Τρία σχόλια έχω να κάνω. Συμφωνώ με την δυνατότητα να μπορεί κανείς να αποσύρεται από τη συμφωνία που έχει κάνει δωρεάν. Εάν όμως έχετε μία οικογένεια τεσσάρων, πέντε ατόμων που ταξιδεύουν και στην περίπτωση ε, αλλαγής σχεδίων ζητείτε 10% καταλαβαίνετε τι κόστος σημαίνει αυτό η οικογένεια. Πιστεύω ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει την αναλλακτική λύση ε, δωρεάν να καταγγέλει ένα τέτοιο είδους συμβόλαιο. Και η συμφωνία, η σχετική, θα πρέπει να συνάπτεται και από τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Και όταν υπάρχει μια τέτοιου είδους αλλαγή στην τιμή, θα πρέπει να έχουν συνενέσει από πριν και οι δύο, και το ταξιδιωτικό ε, πρακτορείο και ο καταναλωτής. Δεύτερη παρατήρηση. Το άρθρο 11.5. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλέπετε κατά το όριο ε, η τρεις νύχτες. Και αν δεν υπάρχει χρονική, ε, χρονικός τέτοιος καθορισμός και αναφέρουμε απλώς 100 ευρώ, θα υπάρχει πρόβλημα και δεν ξέρουμε σε λίγα χρόνια εάν τα 100 ευρώ αρκούν για να καλύψει κανείς τα έξοδα τριών ε, ε, διαμονών, τρεις νύχτες στο ξενοδοχείο. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε για, για τρεις νύχτες. Επίσης, 18 μήνες γιατί την εφαρμογή αυτής της οδηγίας δεν είναι επαρκής χρόνος, διότι αν λάβουμε υπόψη αφενός τις ε, διαδικασίες και το πόσο όλες αυτές τις διαδικασίες επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, διότι όλες οι παρεμφερείς επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να την εφαρμόσουν σωστά αυτή την οδηγία, δεν θα του στάσει ο χρόνος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλέψουμε 24 μήνες για να μπορέσει να εφαρμογεί σωστά ο κανονισμός. Εάν θέλετε, Μπορούμε να συμφωνήσουμε και στους 12, αλλά δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα γίνουν σωστά τα πράγματα από τα κράτη-μέλη. Διότι αφενός εμείς θέλουμε να, να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε και τις διάφορες επιχειρήσεις του κλάδου που πρέπει να ξέρουν με απόλυτη σαφήνεια πώς έχει η κατάσταση. Και πάλι θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή την εξαιρετική του δουλειά. Ευχαριστώ κυρία Βάιλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Πολύ σύντομα θα κάνω τις παρατηρήσεις μου, δεν τη διάβασα όλη την έκθεση. Κύριε Μάιερ. Θα ήταν πολύ πιο απλό ίσως να μας κάνετε μία συνοπτική παρουσίαση για να δούμε τι έχει αλλάξει σε σχέση με το 1990 όσον αφορά την οδηγία, τι γίνεται κατάσταση στη Γερμανία, ίσως και σε άλλες χώρες τι συμβαίνει. Το είπε και η κυρία Μακλάκλιν ότι έγιναν, υπήρξαν κάποιες αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αποτελούν πλέον νομολογία και μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή στην πρότασή της. Στην Γερμανία ξέρω ότι έγιναν τέτοιου είδους πρόσφυγες στο δικαστήριο για την προστασία των καταναλωτών ε, έναντι σε επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν. Επίσης, το δικαίωμα ακύρωσης, το θέμα των ε, πολιτικών προβλημάτων, των φυσικών καταστροφών. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πολλές φορές το ΙΠΕΞ στη Γερμανία εκδίδει διάφορες οδηγίες ταξιδιωτικές, μας λέγει μην πάτε στην τάδε χώρα, στη χύψη ωμέγα χώρα, γιατί είναι δύσκολη πολιτική κατάσταση. Τι είδους επιχείρημα είναι αυτό, είναι σοβαρό εάν κάποιος επικαλεστεί αυτό τον λόγο ε, μπορεί να θεωρήσει ότι το επιχείρημά του είναι ορθό. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα πρέπει να τα εξετάσετε. Ξέρουμε ότι είναι πολύπλοκα τα πράγματα, κάθε νομοθεσία είναι διαφορετική και όντως θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια. Τώρα, θα προλάβουμε πριν από το τέλος της θητείας μας να ψηφίσουμε τη σχετική έκθεση. Είναι Πολύ σημαντικό να την ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Γι' αυτό πείτε μας ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κύριε Μάιερ. Κανένας άλλος συνάδελφος από όσον βλέπω δεν ζήτησε το λόγο. Δίνω αμέσω το λόγο λοιπόν στην Επιτροπή η οποία πρέπει να απαντήσει στις διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν. Υπάρχουν και διάφορα θέματα που ίσως που δεν τέθηκαν εδώ που θα θέλετε να αναφέρετε. Σας καλωσορίζω τον κύριο Ματιάκ, την κυρία Μανφρέντι. Σας δίνω το λόγο και στο τέλος για να ολοκληρώσω θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή Όπως και οι συνάδελφοι του κυρίου Μάιερ συγχαίρει τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Χαιρετίζουμε και συμφωνούμε στην πλειοψηφία του στις τροπολογίες που κατατέθηκαν ώστε να μπορέσει περαιτέρω να διευκρινηθεί το περιεχόμενο της οδηγία. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι θέματα τα οποία μας απασχολούν, κυρίως ο ορισμός του αντικειμενικού στόχου αυτών των προτάσεων. Όπως ξέρετε, θέλουμε να υπάρχουν πάρα πολύ σαφή εξηγήσει για το τι ακριβώς σημαίνει ε, πακέτο διακοπών, μέτρα, ρυθμίσεις που προβλέπονται, μην υπάρχει πρόβλημα του ορισμού και την ορολογία. Είναι πρωταρχικής σημασίας το θέμα στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας της τροπολογίας 29 που με την εισαγωγή του όρου ιδιαίτερος in particular φαίνεται ότι αλλάζει το άρθρο στο οποίο απαριθμούνται διάφορα θέματα που αποτελούν ένα πακέτο με το ότι δεν έχουμε να κάνουμε με διεξοδικό κατάλογο θα πρέπει να προσπαθήσουμε τους ορισμούς της Επιτροπής να τους αποσαφηνίσουμε ώστε να μπορέσουμε αντί να κάνουμε τις λίστες αυτές πολύ διεξοδικές αλλά εντελώς διαφορετικές για τους μεν και για τους δεν, προσπαθήσουμε να κάνουμε μια απλοποίηση και ένα ενασμό εμείς ε, ξέρουμε ότι η δουλειά του κυρίου Μάιερ είναι πολύ δύσκολη, διότι το να μπορέσουμε να βρούμε την ε, μέση λύση και τη χρυσή τομή για όλα αυτά τα είδη ταξιδίων που μπορεί να αγοράσει κανείς είναι δύσκολο και μπορούμε να συνεργαστούμε τον εισηγητή. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω κάποιες ανησυχίες που εκφράστηκαν για αυτές τις περίφημες ε, επικουρικές υπηρεσίες συμπληρωματικά πακέτα και όλα αυτά φέρονται στις τροπολογίες 23 και 36 και συμφωνούμε με την πρόθεση που υπάρχει εκ μέρους του εισηγητού να αποσαφινιστούν κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να είναι και εκτός περιεχομένου οδηγίας αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει οι ορισμοί που θα δώσουμε να είναι σαφείς ώστε να καταλαβαίνουν οι καταναλωτέ, τι συμπεριλαμβάνεται και τι όχι. Θα πρέπει και πάλι να δούμε την σωστή διατύπωση, αλλά και πάλι ε, είμαι υπέρ αυτού το οποίο λέγεται, δηλαδή ό,τι πρέπει να μείνει εκτός οδηγίες να μείνει εκτός. Φερρυπίν, η τροπολογία 68 και ο ορισμός του τι σημαίνει σε περίπτωση ανωτέρας βίας, force majeure, ε, ποιο θα πρέπει να είναι το όριο την ε, υποχρεώσεων του οργανωτή όσον αφορά πόσες νύκτες θα πρέπει να πληρώσει πληρωματικά για τους ταξιδιώτες. Τέτοιου θέματα θα πρέπει να τα δούμε λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έχουμε και αναθεώρηση της οδηγίας φορά τα, ε, δικαιώματα των ταξιδιωτών στον τομέα της αεροναυτιλίας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεκτικοί ώστε να μην υπάρχουν ε, αποκλίνουσες απόψεις και να είναι απολύτως σαφές ποια είναι η ευθύνη του καθενός και κυρίως του υπευθύνου ταξιδίου, αλλά θα πρέπει να δούμε για τις περαιτέρω αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε πώς θα τροποποιηθεί, επαναλαμβάνω, και η οδηγία για τους ταξιδιώτες των αεροπορικών εταιρεών. Όπως είπα και το επαναλαμβάνω για τον φάκελο αυτό όσον αφορά το επίπεδο της εναρμόνισης δεν είμαστε δογματικοί. Εξυπακούεται ότι η Επιτροπή είναι εδώ για να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να μιλούν στα πλαίσια του δυνατού μια κοινή γλώσσα. Επίσης πρέπει να πω ότι ίσως υπάρχουν και, άλλοι, και τομείς που χρειάζονται περισσότερη εναρμόνιση από κάποιους άλλους. Αλλά βεβαίως και εδώ και στο Συμβούλιο εμείς ως διαπραγματευτές θα είμαστε υπέρ του να ευρεθούν πάντα εφικτές και λογικές λύσεις. Σας ευχαριστώ κυρία Μαρφέτη, πάρα πολύ σαφείς απαντήσεις που θα πάτε. Είναι 6 και 25 κύριε Μάιερ. Έχουμε το κοκτέιλ μας περιμένει σε 5 λεφτά. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι θα είστε πάρα πολύ σύντομος. Ευχαριστώ, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω αυτή την προσφορά. Η εναρμόνιση πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Έχουμε έναν οργανωτή ταξιδιών που κάνει το ένα το άλλο και μετά πρέπει να δούμε από ποιο αεροδρόμιο θα φύγει ο ταξιδιώτης, που θα προσγειωθεί όλα αυτά βεβαίως εντός της εσωτερικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι εντός μιας χώρας, διότι πολύ συχνά ένα γραφείο ταξιδίων οργανωμένων πουλά κάτι το οποίο υπάρχει και σε ένα άλλο κράτος μέλος. Ποιο δίκαιο ισχύει, το εθνικό δίκαιο ή πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό είχα προτείνει οι διατάξεις της οδηγίας προστασίας των καταναλωτών να περιληφθεί εδώ, διότι ακριβώς έχουμε συνηθίσει να ρυθμίζουμε με ενιαίο τρόπο εντός της Ευρώπης τα θέματα που τίθενται στις διάφορες χώρες. Αυτά τα είχα πει εξ αρχής, αλλά βεβαίως ή ταξίδια. Όχι σε μια χώρα, αλλά ανάμεσα σε πολλές χώρες. Ακόμη κάτι απευθύνομαι στον κύριο Σμιτ. Δεν επιθυμούμε να είναι οι κυβερνήσεις που να προστατεύουν ε, τους καταναλωτές, αλλά να προστατεύονται από την οδηγία, να προστατεύονται σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι μέρος της συζήτησης που δεν έχουμε ακόμη κλείσει. θέλουμε να δώσουμε δικαιώματα στους επιβάτες, στους καταναλωτές σε σχέση με την αεροπορική εταιρεία ή με τον οργανητή ταξιδίων. Δεν πρόκειται καθόλου για το να δούμε από πού φεύγουμε και πού φθάνουμε, τι θα χρησιμοποιήσουμε, ποιο αεροδρόμιο πρέπει να μεταφερθούν οι ταξιδιώτες να αποζημιωθούν, να στεγαστούν, να δούμε επίσης τι πόσα χρήματα τους δίνουμε για μία διανυκτέρευση. Αυτό δεν εξαρτάται από το μέρος από όπου φεύγουμε ή όπου προσγειωνόμαστε. Καλύτερα μία πλήρης εναρμόνιση. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι πρέπει να έχουμε σαφέστερους ορισμούς και να διαφοροποιήσουμε. Ε, συμφωνώ, αυτό προσπάθησα να κάνω. Αλλά βεβαίως το λίγο χρόνο που είχα τη διάθεσή μου δεν μπόρεσα να κάνω καλύτερα. Περιμένω με ανυπομονησία τις τροπολογίες για να έχουμε ένα κείμενο στο δυνατόν ακριβέστερο και σαφέστερο. Ως προς τα επαγγελματικά ταξίδια είναι μια συμφωνία, μια συμφωνία μεταξύ μιας επιχείρησης και μιας άλλης. Εγώ όταν είμαι βουλευτής κάνω κράτηση επειδή ε, είμαι βουλευτής ιδιωτικά. Μπορώ να αρχίσω ένα ταξίδι επαγγελματικό και να το ολοκληρώσω με τουρισμό να προσθέσω μετά μία εβδομάδα διακοπών. Είναι επαγγελματικό ταξίδι ή ιδιωτικό ταξίδι αυτό. Είμαι πολύ ανοιχτός για τα άλλα σημεία. Να δούμε λοιπόν τι θέση σε ισχύ μετά 18 μήνες. 18 μήνες μετά τη μεταφορά. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμη έξι μήνες αργότερα, ούτω ώστε όλοι οι παράγοντες να μπορέσουν να είναι έτοιμοι. Οι 24 μήνες θα είναι μια κάποια ασφάλεια. Ευχαριστώ σε όλους, ευχαριστώ στους κοιόδης εισηγητές και ευχαριστώ τους συναδέλφους είναι ένα ευρύτατο θέμα όπου υπάρχουν πολλά ε, σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στις διάφορες δυνατότητες. Αυτή είναι η δική μας εργασία μας των νομοθετών. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την εξαίρετη συνεργασία με τους διάφορους συναδέλφους. Πάντως, ε, είχατε πολύ λίγες χρονικές ε, προθεσμίες. Ίσως, ναι, ναι, ακόμη κάτι για να δούμε πότε θα ψηφίσουμε το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Πρώτη ανάγνωση, διότι από ό,τι ακούσαμε από το Συμβούλιο πιθανόν δεν, έχουν ακόμα, ε, δεν έχουμε ακόμα την άποψη του Συμβουλίου. ψηφίζουμε στις 11 Φεβρουαρίου και νομίζω ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές τροπολογίες, πράγμα που είναι καλό και υγιές. Έχουμε λοιπόν 18 Δεκεμβρίου στις 12 την προθεσμία για τις τροπολογίες και στις 22-23 ε, ε, Ιανουαρίου θα εξεταστούν και στην Ολομέλεια του Μαρτίου θα ψηφιστούν. Σας ευχαριστώ όλους. Χαίρομαι λοιπόν να λύσω τη συνεδρία. Δεν μπορώ να δω τι γίνεται έξω, αλλά θα πρέπει να έχουμε ορισμένα ποτά έξω και όλοι ε, σας ε, είσαστε καλεσμένοι. Χαιρετίζω την Λιθουανική ε, Προεδρία εδώ και ελπίζω να έρχεται να πιείτε ένα ποτό μαζί μας και η κυρία Μανφρέντη και οι συνάδελφοι και επίση, οι διερμηνείς που εργάζονται σκληρά είναι καλεσμένοι να πιούν ένα ποτό μαζί μας. Και αύριο το πρωί θα συνεδριάσουμε στι 9. Ελπίζω να είστε σε φόρμα για να ψηφίσουμε στι 9.45. Ευχαριστώ πολύ.